Ladies and gentlemen, Καλώς ήλθατε κυρίες και κύριοι. Μερικές ανακοινώσεις καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι για τις γλώσσες διερμηνίας έχουμε τις γλώσσες των, των τακτικών μελών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ολλανδικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, φιλανδικά, εστονικά, πολωνικά και ρουμανικά έχουμε. Η συνεδρίαση Μετά μεταδίδεται και στο διαδίκτυο. Και θα ήθελα καταρχήν να ξέρω αν έχετε κάποιε παρατηρήσει για την ημερησία διάταξη. Αν όχι, <clears throat> θεωρείτε ότι έχει εγκριθεί η ημερησία διάταξη. Δεύτερο σημείο ανακοινωση του Προέδρου. Απολύτω τίποτα δεν έχουν να σα ανακοινώσω. Και αυτό σημαίνει εξοικονόμηση χρόνου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να καλωσορίσω τους ε, καλεσμένους μου, τον ε, αντιστράτηγο Τον Φανός, τον Γενικό Διευθυντή του Στρατιωτικού Προσωπικού της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Είχαμε και στο παρελθόν επίσημες συναντήσεις, αλλά και άτυπες συναντήσεις. <coughs> Δεν θα σας παρουσιάσω λοιπόν αν κάποιος ενδιαφέρεται, το βιογραφικό του κυρίου Φαν είναι στο φάκελό σας. Στρατηγέ μου. Από ό,τι γνωρίζω, ελπίζω να μην είναι τελευταία μου μας επαφή, λέει ο κύριος Φανός. Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαμοιραζόμαστε την εμπειρία σας μετά από αυτό το διάστημα που είσαστε επικεφαλής της, του στρατιωτικού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να σταθούμε σε ορισμένα ερωτήματα και ιδιαίτερα για τις στρατιωτικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και τη δική σας άποψη καθώς και τις προσδοκίες σας στα θέματα αυτά. Βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή όπου ζητείται από όλους μας να εκφράσουμε την απόψή μας για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλιση και το μέλλον της και εγώ προσκληθεί σε διάφορες συνδιασκέψεις για να λάβω το λόγο για τα θέματα αυτά και είναι χρήσιμο να ξεπεραστούν κάποιες παρεξηγήσεις ή τουλάχιστον έλλειψη κατανόηση που υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών για τα θέματα αυτά. Στατηγέ μου σας δίνω το λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία που έχω να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής σας. Για μένα είναι πάντα ενδιαφέρον να ακούω τα σχόλια των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί και εμείς χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας για να εξασφαλίσουμε ότι θα λειτουργήσουν σωστά τα πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για όλους μας. Εντυπωσιάζομαι επίσης και από τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής σας έχετε συντάξει πολλές εκθέσεις, όπως είναι η έκθεση της κυρίας ε, Γκάμισχ για την ε, ε, στρατιωτική διάσταση των, για την αυτική διάσταση μάλλον της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα για να μπορούμε να βρούμε τον δρόμο προς τον οποίο πρέπει να κινηθούμε. Στη σύντομη μου ενημέρωση εγώ θα ήθελα να σας κάνω κάποιες αρχικές δηλώσεις, να δώσω σύντομες εξηγήσει και ελπίζω ότι θα υπάρξει αρκετό αρκετός χρόνος για ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω για οποιοδήποτε θέμα που άπτεται τη ΣΚΕΠΑ. αλλά στην αρχική μου παρέμβαση θα σταθώ σε ένα γενικό επίπεδο για τα θέματα τα οποία για μένα είναι ζωτικά ως, γενικές, ως γενικές εξελίξεις και τάσεις που αναδύονται. Με έχετε ρωτήσει πώς βλέπω τα θέματα της εξέλιξης της ΚΕΠΑ και της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Το ερώτημά μου άμυνα σε σχέση με τι. Υπάρχουν πολλά έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες που αναφέρονται στις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοκρατία, σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτους δικαίου κτλ. Αν συνοψίσω όλα αυτά τα στοιχεία, ο στόχο μας είναι να εξασφαλίσουμε την ευμάρεια και την ασφάλεια του πληθυσμού μας. Ως ε, στρατιωτικοί και συγγνώμη αν επαναλαμβάνουμε μερικέ φορέ, είμαστε οι πρώτοι που καταλαβαίνουμε ότι όλοι αυτοί οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν μόνο με στρατιωτικά μέσα. Μας λένε πάρα πολύ <clears throat> ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε ποια είναι τα όρια της επίλυσης κρίσεων με στρατιωτικά μέσα. Ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η προστασία της ευμάρειας και η εξασφάλιση της ασφάλειας μόνο με στρατιωτικά μέσα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια συνολική αντιμετώπιση. Όλες οι χώρες σας σχεδόν αναφέρονται στα θέματα αυτά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Εγώ έχω περάσει όλη μου την καριέρα στο ΝΑΤΟ και σε συμμαχίες των ε, εθελοντών, αυτών που θέλουν να λάβουν μέρο σε αυτές τις συμμαχίε, πάντα περίμενα να καταλάβουν και οι διπλωμάτες ότι και αυτοί δεν μπορούν να επιτύχουν μόνοι τους στόχου του χωρίς τη βοήθεια στρατιωτικών δυνάμεων, δυνάμεων διατήρησης της τάξεω, ανθρωπιστικών αποστολών κτλ. Όλα αυτά είναι διαφορετικά εργαλεία και θέλουμε όλα αυτά τα εργαλεία να συναρμόζονται με έναν τρόπο ο οποίο θα είναι συμπληρωματικό και, συγχρονισ... και συγχρονισμένα θα πρέπει να αναπτύσσονται όλα αυτά τα στοιχεία για να επιτευχθεί ο στόχο. Είναι προφανές ότι σε πολλές κρίσεις χρειαζόμαστε στρατιωτικέ ικανότητες γιατί δεν μπορούν να επιληθούν αυτές οι κρίσεις χωρίς χρήση στρατιωτικών μέσων. Επομένω. εγώ πιστεύω ότι το πρώτο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι είναι απαραίτητη μια συνολική αντιμετώπιση και πρέπει να περιέχει και μια σημαντική στρατιωτική συνιστώσα αυτή τη συνολική προσέγγιση. Δεύτερη μου παρατήρηση, η ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωση είναι ακριβώς αυτή η συνολική προσέγγιση. Εντυπωσιάζομαι για το πόσο καλά λειτουργούν όλα αυτά. Ενώ στην αρχή είχαμε πολλές δυσκολίες. Αποφασίσαμε να έχουμε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, έχουμε την ύπατη εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο της Κομισιόν, η οποία είναι επικεφαλής της ε, πολιτικής αυτής. Η εντολή της είναι, όπως γνωρίζετε, ο συντονισμός όλων των εξωτερικών δράσεων και το πράτη Δεν σας λέω ότι είναι κάτι το εύκολο, γιατί υπάρχουν διαφορετικές <clears throat> αντιμετωπίσεις και κουλτούρες και υπηρεσίες και νομικά πλαίσια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αλλά αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι αυτή η προσέγγιση λειτουργεί, ότι οδηγεί σε καλά αποτέλεσματα, όπως στην περίπτωση του κέρατος της Αφρικής και του Σαχέλ. Και οι δυσκολίες του παρελθόντος οφειλόντουσαν σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη πρέποντος συντονισμού, αλλά τώρα αν υπάρξει μια νέα κρίση, η ύπατος εκπρόσωπος είπατε εκπρόσωπο κυρία Άστον καλεί όλους τους εμπλεκόμενους και κινητοποιεί όλα τα εργαλεία τα οποία θα έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο για την επίλυση αυτής της κρίσης και συντονίζουμε <clears throat> τον τρόπο με τον οποίο θα εμπλακούμε έχουμε μια καλύτερη επίγνωση των συνθηκών μπορούμε να συζητήσουμε ποιοι είναι οι επιδιωκόμενοι στόχοι και τα καλύτερα εργαλεία για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς και αυτό από κοινού και συγχρονισμένα. Και πράγματι μπορείτε να θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα θέλετε για οποιαδήποτε κρίση στην οποία μπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περισσότερο από το αριθμητικό άθροισμα των εθνικών προσπαθειών. Έχουμε επίσης και ενδείξεις ότι η στρατιωτική δράση γίνεται πιο αποδοτική και πιο αποτελεσματική με τη συνολική αυτή προσέγγιση. Δεν θα μπω τώρα σε παραδείγματα. Στα ερωτήματά σα είμαι σίγουρο ότι θα αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα περάσω όμω σε μια τρίτη δήλωση. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, γιατί πολλέ φορέ υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις για το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μονάχα μια ήπια δύναμη. Αν έχει κανεί την ισχύ, μπορεί να είναι και ήπιο. Αν είναι ήπιο, αυτό δεν σημαίνει μπορεί να έχει και ισχύ. Εγώ πιστεύω και όλοι θα πρέπει να έχουν αυτή την άποψη. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν αποφασίσει να έχουν μια στρατηγική ασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν συμφωνήσει για τους στόχους και τα εγχειρήματα που θα πρέπει να αναλάβουν οι στρατιωτικές δυνάμεις. Όλα αυτά βρισκόνται μέσα στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ότι ξεκινάμε με ήπιες ενέργειες όπως είναι η υποστήριξη σε ανθρωπιστικές ενέργειες, σε εκένωση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέματα διατήρησης της ειρήνης. Αλλά όταν αυτά πρέπει να γίνουν σε συνθήκες όπου είναι επισφαλής η ειρήνη, τότε θα πρέπει κανείς να δράσει και αυτό σημαίνει χρησιμοποίηση σκληρής δύναμης και όχι ήπιας δύναμης. Έχουμε και την αστυνόμευση της ειρήνης. Πρέπει να υπάρξει αντιπαράθεση, να υπάρξει παρέμβαση μάλλον μεταξύ αντιμαχωμένων πλευρών και επομένως θα πρέπει να έχουμε την ικανότητα να αναλάβουμε τέτοιου είδους στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σε γενικές γραμμές, αν διαβάσετε τα έγγραφά μας, ο στόχος μας θα πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες τις κρίσεις στην άμεση γειτονιά μας, εάν αυτές οι κρίσεις επηρεάζουν αρνητικά και απειλούν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι μια έγκυρη για μένα προσέγγιση και εγώ συμφωνώ με αυτούς που λένε ναι, μα αλλά υπάρχει και το ΝΑΤΟ. Υπάρχει το ΝΑΤΟ, αλλά υπάρχουν παρόλα αυτά κάποιες κρίσεις όπου το ΝΑΤΟ δεν θέτει το θέμα ούτε καν στην ημερησία διαταξή του. Και ίσως το μέλλον θα γίνει διαφορετικό. Θα είναι πιο έντονο αυτό γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε για τους δικούς στρατηγικούς λόγους έχουν εστιάσει την προσοχή τους στην λεκάνη του ειρηνικού. Πάρα πολλέ από τις κρίσεις όμως που αντιμετωπίζουμε δεν ενδιαφέρουν άμεσα το ΝΑΤΟ, η Σομαλία, το ΝΑΤΟ, το Κονγκό, ο Νίγηρας, η Λιβύα, η Λιβύη. Υπάρχουν λοιπόν ε, μεγάλα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία διακυβεύονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τέλος, να αναφερθώ στις στρατιωτικές ικανότητες και την ανάπτυξή τους. Και εδώ θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επικαλύπτεται με τον ΝΑΤΟ. Η αρχή μας είναι ότι διευκολύνουμε, διευκολύνουμε και η τορικό προσωπικό και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας υποστηρίζει τη δημιουργία των ικανοτήτων που χρειαζόμαστε αλλά αυτές οι ικανότητες στρατιωτικέ είναι πάντα στα χέρια των κρατών μελών και μπορούν τα κρατημέλη να αποφασίσουν να θα χρησιμοποιήσουν αυτέ τις ικανότητες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, τις ε, συμμαχίες για συγκεκριμένες ενέργειες. Επομένως, θα πανούμε προσπάθειες για να μπορούμε να έχουμε μια στρατιωτική ικανότητα και αυτό έμεσα ενισχύει και το ΝΑΤΟ. Πέμπτη παρατήρηση. Αν θέλουμε οι στρατιωτικοί να είναι τμήμα μια συνολική προσέγγιση, <clears throat> θα πρέπει να έχουν επαρκεί δυνατότητε σχεδίαση για να μπορέσουν να καταστρώνουν σχέδια που κινούν με του πολιτικού του μη στρατιωτικού εταίρου μα. Όλοι οι μη στρατιωτικοί συνεργάτε μου και εταίροι μου έχουν την ικανότητα σχεδιασμού και μπορούν και με στρατιωτικούς όρους να μπουν στις λεπτομέρειες επιχειρησιακών σχεδίων ο συνάδελφός μου από τις μη στρατιωτικές ενέργειες που ασχολείται με τις αποστολές αστυνομικού χαρακτήρα χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια ορολογία με μένα και φυσικά έχει και τη δική του αυτόνομη ικανότητα σχεδιασμού. Θα ήταν πολύ παράξενο να πούμε ότι είναι συνολική προσέγγιση η ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μόνο εργαλείο σχεδίασης μάλλον το μόνο ουσιαστικό εργαλείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στρατιωτικοί να μην έχουν αυτόνομη ικανότητα σχεδίαση. γιατί αυτό θα οδηγούσε σε καθυστέρηση. Και ενώ η στρατιωτική είναι το πιο γρήγορο εργαλείο αντίδραση σε επίπεδο τακτική δράση στι Βρυξέλλες πολλέ φορές παρεμβαίνουν καθυστερήσει. Όλα αυτά μπορεί να είναι χρήσιμα και θετικά σε αποστολές διατήρησης ειρήνης, αλλά για πιο μικρές και ευέλικτες ενέργειες όπως αυτή στη Σομαλία, δεν έχει νόημα να κινητοποιήσουμε όλα αυτά τα κέντρα σχεδίασης που δεν είναι απαραίτητα για μια τέτοια μορφή σχεδίασης. Πρέπει όμως να ζητήσουμε πάντα από μια χώρα μέλος να αναλάβει τη σχεδίαση και την ηγεσία της δράσης. Για τη Σομαλία ήταν η Ισπανία στη Μαδρίτη αν θέλουμε να κάνουμε μια αστυνομική ενέργεια, τότε ο σχεδιασμός θα γίνει εδώ, στις Βρυξέλλες. Και εδώ δεν έχουμε την βέλτιστη μορφή σχεδίασης και να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες συνέργειες. Είναι πολλά λοιπόν τα οποία πρέπει να γίνουν από κοινού, η επιμελητία, η εξασφάλιση των υποδομών, η ιατροφαρμακευτική υποστήριξη, η προστασία των δυνάμεων. Θα ήταν πολύ χρήσιμο λοιπόν αν το δικό μου προσωπικό να έχει τους σχεδιαστές οι οποίοι μαζί με τους ε, σχεδιαστές από την πολιτική πτυχή να μπορέσουν να εργαστούν από εκείνου για να έχουμε αυτή την πλήρη συνολική στρατηγική. Δεν σας ζητώ να έχουμε ένα τεράστιο επιτελείο, δεν θέλω να διπλασιάσω τις δυνάμεις που υπάρχουν και να επικαλυφθώ με τον ΝΑΤΟ. Απλώς θα πρέπει να έχουμε το απαραίτητο προσωπικό. Με 20 σχεδιαστές εγώ θα μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Περνώ στο επόμενο σημείο. Σε ένα πολύπλοκο πλαίσιο. Και ας είμαστε σαφείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πολύπλοκος χώρος. Πολλά νομικά πλαίσια, πολλές υπηρεσίες, <clears throat> πολλές ε, και πολύμορφες διαδικασίες λήψης απόφασης. Σε αυτό το πολύπλοκο πλαίσιο, για μένα, η απλότητα είναι το καλύτερο κριτήριο για τη σωστή οργάνωση. Αν από αυτήν την στρατιωτική προσέγγιση και οπτική γωνία. Δω πώς οργανώνονται τα πράγματα στα κράτη-μέλη. Με δύο εξαιρέσεις, όλα τα κράτη-μέλη έχουν ένα Υπουργείο Άμυνας, πέραν του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχουμε ένα επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος έχει στρατιωτικό προσωπικό για να τον υποστηρίξει, γενικό επιτελείο, αμυντικό επιτελείο κτλ. με διάφορα ονόματα πάντα Όλα αυτά είναι απλά, τα καταλαβαίνουμε όλοι. Εγώ πρέπει να συνεργαστώ με αυτές τις δομές. Χρησιμοποιώ τις πολιτικές ε, διαδικασίες και δομές. Ε, φυσικά καταφεύγω στην Βαρονέσα Άστον. Εγώ είμαι το στρατιωτικό της Μπράτσου και εργάζομαι και στα πλαίσια της Στρατιωτική Επιτροπής τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχω και το, το στρατιωτικό προσωπικό που εργάζεται σε επίπεδο επιτέλειων. Γι' αυτό η συνεργασία με τα κράτη-μέλη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο το καταλαβαίνουν όλοι, είναι πιο εύκολη η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ μας και η αρμοδιότητες είναι σαφείς. Οποιαδήποτε όταν βγαίνουμε από αυτό το πλαίσιο, τότε τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα στη συνέχεια. Γιατί θα φύγουμε από το πλαίσιο το οποίο γνωρίζουμε μέσα στην ε, εθνική και ευρωπαϊκή διάταξη πραγμάτων. Σήμερα δεν είναι να το αποκριθεί Στι φιλοδοξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα περισσότερα κρατημέλη συμφωνούν προ τούτο. Εάν δεν ρίξουμε μια ματιά όσα αποφάσισαμε το 2008, δηλαδή να έχουμε βασικό στόχο ορόσημο το 2010 και κατόπιν επί μια διετία να προσπαθήσουμε να πετύχουμε το στόχο, ε, διαπιστώνουμε ότι ποτέ δεν το πετύχαμε. Από δε το 2010 ουσιαστικά είμαστε σε ελεύθερη πτώση γιατί έχουμε δραματικές περικοπές σε όλα τα κράτη-μέλη και πάμε στο 15-20% περικοπή και ίσως ε, σε μερικά κράτη παραπάνω, για μερικά κράτη-μέλη δεν μπορέσαν να συντονιστούν ε, με τον ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το τι θα περικόψουν. Σχεδόν παντού οι περικοπές γίνονται επί τη βάση εθνικών κριτηρίων. Και, και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επομένως ε, αυτή τη στιγμή τώρα βρισκόμαστε σε κάποια μηχανία, δεν ξέρουμε πού είναι τα πράγματα, γιατί όντω αντιλούμε πληροφορίε, αλλά ε, οι πληροφορίε αυτέ δεν είναι τέτοιε που να έχουμε όλο το ψηφοδοτό, κάτι το, οποίο ε, φέρνει κάποιο είδου φόβο. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Είναι πολύ συγκρατημένοι στόχοι μα. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε κάποια απειλή από την άμεση γειτονιά μα. Ρίξτε μια ματιά εκεί ε, σε το τι κρίση σοβούν εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τις επιλύσουμε. Άρα, τι μπορεί να απαντήσει κανείς σε αυτό το οποίο ρωτήσατε, ποιο είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Αμήνης. Δεν μπορώ παρά να πω ότι θα έπρεπε να είναι το μέλλον λαμπρό. Κρίμα που θα πρέπει να αποχωρήσω γιατί μπορώ να σκεφτώ λόγους που συντείνουν, που κατατείνουν μόνο στην περαιτέρω βελτίωση. Και βεβαίω δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε την δύναμη, την ισχύ, το πόσο σημαντικό είναι το ΝΑΤΟ για κάποιο είδου υψηλή ένταση σύγκρουση όπου έχει το περίφημο άρθρο 5 το οποίο άρθρο 5 μπορεί να υπάρχει μόνο για το ΝΑΤΟ και αυτό χρειάζεται γιατί χρειαζόμαστε να είναι μέσα στο παιχνίδι η ΙΠΑ και σε σχέση, σε σύνδεση με το ΝΑΤΟ και χάρη σε αυτό μπορώ να οργανώσω κάποιες τέτοιες επιχειρήσεις γιατί τη διαλειτουργικότητα, την προτυποποίηση, όλα αυτά τα φροντίζει το ΝΑΤΟ και εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε κανένα είδους ε, ε, αναπαραγωγή, επικάλυψη γιατί τα κράτη-μέλη ε, έχουν πρόσβαση σε αυτές τις δομές του ΝΑΤΟ. Πολλά παραδείγματα έχουμε που κατατείνουν στο ότι θα πρέπει να υπάρχει συνολική εμπλοκή και χρειάζεται τελικά και πολιτική συνιστόσα όσοι συγγνώμη είστε, είστε θετικοί στο Δυτικό Βραχίωνο. Τώρα, ποιο είναι το επόμενο ορόσημο και για ποιο λόγο έχετε εδώ διάφορα θέματα να συζητήσετε στην ημέρα σε διάταξη. Και βέβαια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του τέλους του ενεστώτος έτους και είναι γι' αυτό πάρα πολύ σημαντικό κανείς να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί να αξιολογήσει, να αξιοποιήσει την, αυτό το Συμβούλιο. Τώρα από πλευρά στρατιωτική. Τι μπορούμε να περιμένουμε από εκείνο το Συμβούλιο. Μπορούμε να πούμε κάποιες γενικόλογες παρατηρήσεις σχετικά. Εγώ θα ήθελα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να αναγνωρίσουν το πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ω στρατιωτικό και αυτό σε σχέση με κάποια προσέγγιση σφαιρική. Δεύτερον, να τονίσουν αυτοί όλοι ε, την ε, φιλοδοξία τη Ένωση που ισχύει ακόμα σαν βασική φιλοσοφία. Και άρα επομένω θα πρέπει να είμαστε στη θέση να να διεκπεραιώσουμε, να επιλύσουμε προβλήματα περιφερειακά και κρίσεις τέτοιες, αν δεν μπορεί κάποιος άλλος. Τρίτον, για να γίνουν τέτοια, τέτοια θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους έστω και μετρίου επίπεδου επιχειρησιακή δυνατότητα και επίσης να γνωρίσουν ότι υπάρχει μεταξύ φιλοδοξίας και ικανότητος και δυνατοτήτων τεράστιο κενό σήμερα και άρα θα πρέπει και εμείς τώρα να επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας ούτως ώστε να αναπτύξουμε τις δυνατότητες ε, να αναπτύξουμε την, ε, όπως λέει το ΝΑΤΟ, την, την, τον στρατιωτικό, τον αμυντικό σχεδιασμό και οπότε τον Δεκέμβριο ε, τα πράγματα να έχουν, κάνει, να έχουν προχωρήσει λίγο το Δεκέμβριο που θα συναντηθούν αυτοί όλοι εκείνοι, η αρχή κρατική κυβέρνηση και επίση κατά πέμπτον να γίνει κατανοητό ότι περαιτέρω περικοπέ στον αμυντικό προπολογισμό θα είναι κάτι τραγικό για την προστασία της ευημερία της και για την ασφάλεια. Και οπότε να αναγνωριστεί ότι είμαστε πλέον στα, στα όρια του παραδέκτου σύμβρα τις περικοπές και γι' αυτό θα πρέπει η ευημερία και η ασφάλεια να αποτελέσουν αντικείμενο επένδυσης. Σε σχέση με όλα αυτά τώρα, αυτό που προσβεύω είναι και οι υπουργοί, αλλά και οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων να αναλογιστούν το πώς με τον δεδομένο προπολογισμό είναι πιο αποτελεσματική και να σκεφτούν το ότι οι αμυντικές πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Δεν είναι για μια στόχη αλλά ρωτάω το, το, επιτελείο μου. πώς άλλο θα χρειαζόταν τόσο να υπάρχουν κάποιε τέτοιε πρωτοβουλίε, να υπάρχει συντονισμό. Και έτσι ουσιαστικά θα εξοικονομήσουμε δαπάνε. Κατά πρώτον αποταμιεύουμε με αυτές τις περικοπές και δεύτερον επενδύουμε. Οπότε αν κάτσουμε και δούμε όλες τις οικονομίες που έχουμε κάνει μιλάμε για ε, εξοικονόμηση 200-300 εκατομμυρίων. Κάτι το οποίο είναι υπέροχο γιατί 300 εκατομμύρια το χρόνο είναι ένα πάρα πολύ όμορφο ποσό. Επίσης, τους λέω στο προσωπικό για κοιτάξτε στο ίντερνετ Πώ ήταν όλε μαζί οι περικοπέ στην Ένωση. Διαπιστώνετε ότι μιλούμε για 30 δι. 100 φορές δηλαδή παραπάνω περικόψαμε από όσο είναι η ενδυνάμει εξοικονομήσεις. Ναι, αλλά πρώτα κανεί πρέπει να επενδύσει. Να, ένα απλό παράδειγμα. Πυρωτική κατάρτιση. Όλοι μαζί. Και όχι ο καθένα τη, τη δική του κατάρτιση. Όμω πρώτα θα πρέπει να γίνει επένδυση. Ας πούμε οι Γάλλοι να βελτιώσουν τις σωτικέ σχολέ, τη Σίτρα, τις αντίστοιχες σχολές, πριν γίνει αυτή η συντονισμένη προσπάθεια. Γιατί η χώρα που θα αναλάβει την κατάρτιση θα πρέπει για τους πιλότους, ας πούμε, να εκταμιεύσει κάποια ποσά. Άρα, εξοικονόμηση, αφενός, αφετέρου όμως, εκατονταπλάσιες περικοπές από τις εξοικονομήσεις. Αυτό γίνεται. Τώρα, παραπέρα από τα θέματα του χαρτοφυλακίου μου, του ορμοδιοτήτων μου, ελπίζω ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα αναγνωρίσουν ότι όπως και για όλους τους κλάδους και η αμυντική βιομηχανία είναι πάρα πολύ σημαντική για την απασχόληση αλλά και για την προστασία των, ανθρωπι... των ευρωπαϊκών αξιών. Και ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος. Εγώ σας ευχαριστώ. Είχα και εγώ δύο ερωτήσεις προς τον στρατηγό. Πρώτα πρώτα. Για τις προσδοκίες σας, για τις αντισυκορυφίες και η δεύτερη ερώτηση. Τι θα γίνει με την ευφύ άμυνα εν αυτών των περικοπών. Αλλά με καλύψατε και θα δώσω τώρα τη σκητάλη στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Γκάλερ, Κοπά, Φανόρντεν, κάτω. Συγγνώμη, συγγνώμη. Εν δεν ε, παστώ το όνομά σα. Πολύ, πολύ συνάδελφοι στο λόγο. Άρα, τώρα θα ήθελα να σα ερωτήσω Μήπω μπορείτε να μιλήσετε το πολύ δύο λεπτά. Για να ακούσουμε και τι απαντήσει του στρατηγού. Κύριε Γκάλ, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ. Και με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα τις ε, επεξηγήσεις σας. Θα είχα και εγώ να σας κάνω την ερώτηση που εν μέρει απαντήσατε. Τι αναμένετε, τι προσδοκάτε από την Σύνοδο. Το ξεκαθαρίσατε αυτό. Θεωρώ ότι θα το παρουσιάσετε αυτό με την κατάλληλη μορφή και στις ε, ανάλογες επιτροπές, στα ανάλογα φόρα. Νομίζω ότι και μόνο ο αριθμός ε, των περικοπών που αποτελεί το εκατονταπλάσιο των όσων έχουν περικοπεί στα κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην αγγλική καμπίνα, ρωτάει ο Πρόεδρος. Είναι ακόμα στην Ένωση η Αγγλία. Ναι, έχετε πολλές άλλες γλώσσες να επιλέξετε, λέει ο Πρόεδρος. Uh, Τώρα εντάξει, μάλιστα. Δεν θα μιλήσω αγγλικά για να δουλέψει και η αγγλική καμπίνα, λέει ο κύριος Γκάλερ. Όλα καλά τώρα, επιλύθηκε το πρόβλημα. Πορτογαλικά, όχι, πορτογαλικά δεν θα μιλήσω. Θα μιλήσω αγγλικά. Υποθέτω ότι στο Συμβούλιο οι θύνοντες γνωρίζουν τι θα πρέπει να γίνει και τι χρειαζόμαστε. Δεν πρόκειται να κάνουμε εικασίες ασφαλώς στην παρούσα φάση για το τι θα σκεφτούν. Απαντήσατε λοιπόν αυτή την ερώτηση ουσιαστικά πριν σας τη θέσω. Αναρωτιέμαι σε ό,τι αφορά την διαθεσμική συνεργασία στο εσωτερικό της Ένωσης. Σε τι βαθμό μπορεί να συνδράμει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάπτυξη του δυναμικού. Έχουν πολλά κονδύλια για πολλούς σκοπούς. Και πολλές ε, είναι οι δυνατότητες ε, που μπορεί να ωφελήσουν και τον ε, πολιτικό τομέα και να έχουν και εφαρμογές στον στρατιωτικό τομέα. Αναρωτιέμαι, όπως εξηγήσατε, δεν υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις σε ό,τι αφορά το έργο μας με τον ΝΑΤΟ. Φυσικά αυτό πρέπει να κάποιο συντονισμό με τον ΝΑΤΟ για να αποφευθούν ενδεχόμενες επικαλύψεις. Και επίσης σημειώνουμε ότι οι Αμερικανοί φίλοι μας συχνά μας λένε ότι θα πρέπει να φροντίσουμε πρώτα τα του δικού μας οίκου. Ερωτώ, υπάρχει λοιπόν κάποιος προηγμένος συντονισμός προκειμένου να γνωρίσουμε τι, μας, ε, τι θα μας φέρει το μέλλον σε ό,τι αφορά ενδεχόμενες κρίσεις στη Γουινέα, για παράδειγμα, στον κόλπο της Γουινέας ενδεχομένως να ανακύψει κάτι συντόμως. Πρόκειται για ένα τομέα συντονισμού με τον ΝΑΤΟ, ενδεχομένως. Αυτό το, ανα... το αναφέρω ενδεικτικά ως παράδειγμα. Αυτά στην παρούσα φάση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Κοπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Όντως, προσπαθήσατε να μας δώσετε μία επισκόπηση της κατάστασης και να καλύψετε όλα τα θέματα τα οποία ενδεχομένω θα σας ε, θέταμε ως ερωτήσεις. Δύο ζητήματα σε ό,τι αφορά καταρχάς... Ε, σε ό,τι αφορά τις ε, περικοπές βρισκόμαστε σε, σε μια τέτοια περίοδο περικοπών πέρα από το να μιλάμε για την ε, άμυνα, για την κοινή διαχείριση και την κοινή δαπάνη κονδυλίων που όντως έχουν τη θέση τους ε, στη συζήτησή μας. Ε, υπάρχει κάποια νέα στρατηγική από πλευρά σας για το νέο αυτό οικονομικό περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε και ύστερα κατά δεύτερον μας δίνετε μια ιδεαλιστική, αν θέλετε, μια ιδανική εικόνα για τη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Ενώ υπάρχουν ακόμα επιχειρήσεις όπου η συνύπαρξη δεν είναι αυτονόητη και εύκολη. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας παρουσιάσετε και την δύσκολη πλευρά της ε, συνεργασίας αυτής στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και μια τρίτη ερώτηση για τις απειλές στον κύβερνο χώρο. Τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Άμυνα για αυτές. Ευχαριστώ. Κρόνμπεργκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε αυτό το pooling and sharing στην κοινή ε, δαπάνη κονδυλίων. Τα αριθμητικά στοιχεία που μας δώσατε είναι πάρα πολύ ε, θετικά και η ιδέα να ξεκονομήσουμε 30 δισεκατομμύρια και 200 εκατομμύρια στο pooling and sharing. Αλλά Πώς αντιμετωπίζουν τα κρατημέλη αυτό το pooling and sharing, γιατί από ό,τι κατάλαβα το βασικό πρόβλημα είναι η εμπιστοσύνη. Πώς θα οικοδομηθεί αυτή η εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει κοινή οργάνωση, να υπάρχει αυτό το pooling and sharing. Δεύτερη ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση στο Μάλι. Πότε θα καταστεί λειτουργική και πόσοι στρατιώτες θα αποσταλούν και πώς έχει η κατάσταση ε, σε ό,τι αφορά την ασφάλειά τους και τι, ποιες ανάγκες υπάρχουν. Ευχαριστώ, ο κύριος Πανόρντεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και στρατηγέ, πάντα σας ακούμε με ιδιαίτερη χαρά στα αγγλικά, λέμε. Και λέμε ότι καλό είναι να τα ακούμε από το, από το στόμα του αλόγου. για να ξέρουμε τι είναι αξιόπιστο, να τα ακούμε τα πράγματα από την πηγή τους. Ξέρω ότι συχνά μας αρέσει να σκεφτόμαστε ότι οι ΕΠΑ κινούνται προς την Ασία και ότι αυτό αποτελεί δικαιολογία και για την Ευρώπη. Αυτό δεν ισχύει πάντα ασφαλώς. Αυτά που λένε πάντα οι ΙΠΑ και έλεγανε πάντα είναι ότι θέλουν να ε, μοιραστούν το φορτίο της εργασίας με τους Ευρωπαίους συμμάχους. Αυτό το λένε τα τελευταία 50-60 χρόνια. Δυστυχώς ε, οι ΕΠΑ συχνά λένε επίσης ότι η Ευρώπη κάνει τα, τη δική της οργάνωση, Τη, τη δική της οργάνωση. σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τον ΝΑΤΟ και πάλι τα ίδια κρατή μέλη κάθονται γύρω από μια στρογγυλή τράπεζα και είναι απόλυτο ανόητο το ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ε, συντονισμού, γιατί οι εκπρόσωποι είναι ουσιαστικά εκπρόσωποι των ίδιων χωρών λίγο πολύ και συνεδριάζουν και στην ίδια χώρα και στην ίδια πόλη. Και σε κάποια φάση κάθε κράτος ε, μέλος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει συμμετάσχει σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Γιατί να μην λαμβάνει λοιπόν όλα αυτά χώρα στο ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. ένα λόγο. Η απλότητα των υποδομών που αναφέρατε είναι οι ίδιες υποδομές που έχει το ΝΑΤΟ τα τελευταία 50 χρόνια. Και τις έχει ουσιαστικά α, επαναλάβει, τις έχει ξαναχτίσει η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την το στρατιωτικό επιτελείο, τη στρατιωτική επιτροπή, τους εκπροσώπους που ε, συνέρχονται κάθε μέρα σχεδόν. Είναι ακριβώς η ίδια δομή με το στρατιωτικό επιτελείο. Δεν πρόκειται για τίποτα το καινοτόμο και θα πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να βρει ε, μια καλή δικαιολογία για την ΚΕΠΑ, πέρα από την πραγματικό σκοπό που είναι ασφαλώς να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση μια παγκόσμια συνιστόσα. Και τώρα αναφέρεται η συνεκτική προσέγγιση που χρησιμοποιεί διάφορες ε, δικαιολογίες και τώρα αναφέρεται λοιπόν αυτή η συνεκτική προσέγγιση. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε μία επιχείρηση στα θετική των τελευταίων δέκα ετών που δεν έχουν περιλάβει ε, και ένα σχέδιο πολιτικό, πολιτικού σκέλους. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα το καινούργιο σε αυτή τη συνεκτική προσέγγιση και για το, ο λόγος για τον οποίο κάποιες ε, κρίσεις ε, δεν είναι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ είναι επειδή το έχουν επιλέξει κάποια κράτη-μέλη γιατί προτιμούν να το διαπραγματευτούν κάπου αλλού το θέμα αυτό για να δώσουν αρμοδιότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέσσερις ερωτήσει τώρα, ε, στρατηγέ. Λέτε ότι δεν επαναλαμβάνουμε και δεν ε, ε, κάνουμε διπλό έργο σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Τι δυνατότητες, δυνατότητες δημιουργούνται που δεν υπήρχαν πριν για τα κράτη-μέλη και που θεωρείτε ότι είναι σημαντικές σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ. Κατά δεύτερον, Ποιο είναι το πιο σημαντικό επόμενο βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προωθήσει τον ρόλο της ε, στην άμυνα. Τρίτον, πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει προϋπολογισμό για την άμυνα. Και τέταρτον, δεδομένου το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί αυτό που αποκαλώ ανθρωπιστική βοήθεια, ανθρωπιστική αρρωγή για δικαιολογία πολλών όσων κάνει, χρησιμοποιεί ευρέω τον όρο αυτό, θέλετε κάποια στοιχεία του προϋπολογισμού για την ανάπτυξη και την, ε, να χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, επόμενος ομιλητής. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα με την ε, ιδεαλιστική σας προσέγγιση. Το βασικό σας μήνυμα θεωρώ είναι ότι υπάρχει μεγάλο κενό μεταξύ των ε, φιλοδοξιών και των ικανοτήτων μας, των δυνατοτήτων μας. Α, είπατε ότι περαιτέρω περικοπές θα αποβούν μοιραίες, θα είναι καταστροφικές. Φυσικά υπάρχουν κάποιες χώρες που δεν έχουν υποκύψει στις πιέσεις αυτής. Εγώ εκπροσωπώ την Εστονία που εξακολουθεί να δαπανά 2% για την εθνική άμυνα, αλλά είμαστε μικρή χώρα και ουσιαστικά ηθική υποστήριξη και παρέχουμε. Μας υπενθυμίζεται το μήνυμα του Υπουργού Άμυνας και της Πολωνίας την προηγούμενη εβδομάδα που είπε ότι αυτό που συνέβη πριν από τέσσερα χρόνια στον χρηματοοικονομικό τομέα ενδεχομένως να ε, επαναληφθεί στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, γιατί δεν είμαστε προετοιμασμένοι, δεν έχουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς, δεν έχουμε τους απαραίτητους πόρους για να το παρεμποδίσουμε. Αυτό αποτελεί μια κοινή ανησυχία. Η ερώτηση λοιπόν που έχω να σας απευθύνω, όπως και ο συνάδελφος ε, κυρία Κόπα, για τον τομέα της, ε, του κυβερνοχώρου και τις σχετικές απειλές που εμφανίζονται. Πόσο σοβαρές θεωρείτε ότι είναι αυτές οι απειλές ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, θα μπορούσαμε να θέσουμε κάποια ελάχιστα πρότυπα, κάποιες ε, ελάχιστες προδιαγραφές για την υποχρέωση αναφοράς και συντονισμού και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις κρίσεις στον τομέα αυτό, στον κυβερνοχώρο. Αμφιβάλλω κατά πόσο είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι στον, ε, στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Αφοκλέους. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και βέβαια για τα μηνύματα τα οποία έχετε δώσει σήμερα. Εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνηθίζουμε να επαναλαμβάνουμε μία αρχή ότι στον χώρο μας δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική άμυνα και ασφάλεια. αναζητείτε και είναι ερώτημα εάν θα καταφέρουμε και περιορίζουμε σε αυτό, να υπάρξει κοινή άμυνα και ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική μου ερώτηση είναι καθαρά πολιτική και όχι τεχνική, τεχνοκρατική. Εάν με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν με βάση τις οδηγίες, τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή έχουμε μια νομιμοποιημένη επέμβαση θα μπορούσατε με τα σημερινά μέσα να έχετε αποτελεσματική παρουσία και να φέρετε την ειρήνη. Παραδείγματο χάρη, φέρνω δύο παραδείγματα σήμερα στο Μαλί, στη Συρία, όπου έχουμε αιματοχυσίε και βλέπουμε να σκοτώνονται χιλιάδε ανθρώποι, αλλά η ουσιαστική παρέμβαση πρακτικά να μην γίνεται. Και ένα επιμέρους ερώτημα και κλείνω. Αν φτάσουμε κάποτε οραματικά, λέω, στην κοινή εξωτερική πολιτική άμυνα και ασφάλεια που το εύχομαι τουλάχιστον εγώ να υπάρχει κοινή ενιαία πολιτική και για λόγους πολιτικής και για λόγους οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια θα είναι η σχέση με το ΝΑΤΟ. Θα είναι ανταγωνιστική αυτή η σχέση. Θα είναι παραγωγική. Εσείς έχετε γνώση στρατιωτική και εμπειρία και νομίζω θα μας φωτίσετε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ κύριε Γκόμις. Ευχαριστώ. Στρατηγέ, την προηγούμενη Κυριακή η... ένα πρόγραμμα στην Πορτογαλική τηλεόραση γνωστό ως Prime Time που παρουσιάζει τα θετικά και τα αρνητικά σε διάφορα πολιτικά θέματα είχε ένα εξέχον πάνελ από αρχηγούς του στρατού, του ναυτικού, αεροπορίας, αντιτρομοκρατικές ε, δυνάμεις από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Πορτογαλία και υπήρχαν πολύ οργισμένες δηλώσεις κατά της Ευρώπης λόγω των, των περικοπών που γίνονται στις ε, ένοπλες δυνάμεις μας λόγω της λιτότητος. Φυσικά εδώ δεν είναι η ευθύνη μοναχά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και της κυβερνήσεως με τον τρόπο που εφαρμόζει αυτές τις ε, περικοπές χωρίς να μπορεί να τις εξηγήσει στους ανώτατους στρατιωτικούς. Αλλά αναρωτιέμαι, ποια είναι η σχέση που δημιουργεί η Στρατιωτική Επιτροπή με τα γενικά επιτελεία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατανοούν καλύτερα τι είναι αυτά που προσπαθεί να επιτύχει η Ευρώπη μέσα στην κοινή εξωτερική πολιτική ε, και η πολιτική ασφάλειας. Υπήρξαν πολλά χαζά σχόλια που δείχνουν ότι υπάρχει άγνοια αυτής της πολιτικής και υπάρχει μια δυσκολία στο να κατανοήσουν ότι οι εθνικές στρατιωτικές ικανότητες θα ενισχυόντουσαν εάν τις έθετε το κάθε κράτος πιο συχνά στη διάθεση της ΚΕΠΑ. Και ένας από για τους οποίους δεν λαμβάνει χώρα αυτό είναι το θέμα της χρηματοδότησης αυτών των αποστολών της ΚΕΠΑ. Η εκπαιδευτική αποστολή για το Μαλί είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να μπορέσουμε να εστιάσουμε καλύτερα την αντίληψη των πολιτικών ηγετών μας στο, στην ανάγκη να υπάρξει κοινή χρηματοδότηση των αποστολών της ΚΕΠΑ, ώστε χώρες φτωχές όπως η δική μου χώρα, η Πορτογαλία που έχει δυνάμεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια κρίση όπως η κρίση του Μάλι, να χρησιμοποιηθούν πράγματι. Γιατί όπως είναι αυτή η κατάσταση και αυτοί που δεν στέλνουν στρατεύματα εξακολουθούν να πληρώνουν. Γιατί δεν τίθεται λοιπόν σε συζήτηση αυτό από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και όχι μόνο τους στρατιωτικούς αρχηγούς. και για, το, για την κυβερνοασφάλεια. Στη δική μου χώρα δεν υπάρχει καν κέντρο κρίσης που να αντιμετωπίζει τέτοιες ε, κυβερνοεπιθέσεις. Μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μία πλήρη κάλυψη όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρισίμων υποδομών της, γιατί ο πιο αδύναμος κρίκος είναι από εκεί που θα μπορέσει να ευδοκιμήσει η επίθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όσα μας είπατε κύριε Στρατηγέ. Όπως και ο συνάδελφος εδώ, ο Σιόνομο, μου, για αυτό το θέμα της ε, επικάλυψης έχω πρόβλημα στο στο Λονδίνο. Έχουμε τις ΝΑΦΟΡ που είναι 100 μέτρα ε, μετά από την ε, Ατλαντική ασπίδα του ΝΑΤΟ. Και οπότε τι γίνεται. Έχουμε αυτές τις περικοπές και παρόλα που θα έχουμε αυτές τις επικαλύψεις. Αυτό δεν εξυπηρετεί κανένα. Έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις. Πρώτα-πρώτα μας αναφέρατε κάτι σε σχέση με τα συμφέροντα της Ένωσης που επαπειλούνται. Για πέστε μας παρακαλώ. Πότε γίναμε κράτος ως Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εγώ οπότε ξέρω Μιλούμε για εθνικά συμφέροντα εν προκειμένου και αυτό και με προβληματίζει αυτό που είπατε. Επίσης, για την έκθεση Ντονζό, ξέρουμε ότι γίνονται συζητήσεις όσον αφορά την εμπλοκή σε κάποιο είδους ε, σύγκρουση υψηλής έντασης που εγώ το καταβαίνω ως πόλεμο. Εσείς υπό ποιες περιστάσεις θέλετε να, να, να μπείτε σε πόλεμο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιος, θα πιο το εγκρίνει αυτό, ποιος το συμβουλεύει αυτό. Επίσης μιλάτε για αυτές τις ε, πρωτοβουλίες όπως η πιλωτική κατάρτιση, η κοινή κατάρτιση. Και πότε εσείς περιμένετε όλα αυτά να καταλήξουν σε κάποιο είδους κοινές ένοπλες δυνάμεις. Και σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το εξής. Εσείς έχετε μοναδική γνώση, αλλά και πάρα πολύ εκτεταμένη εμπειρία από τα σταθιωτικά πράγματα. Ξέρετε τη διεθνή συγκυρία και επίσης ε, διάβασα το βιογραφικό σας και επίσης έχω εξοικειωθεί, ξέρω καλά, τη διαδρομή σας, τα διδρομία σας, οπότε ως εκτεσθέσιό σας κάνετε πάρα πολλές αποστολές στο Αφγανιστάν, στα Βαλκάνια επίσης. Και ξέρετε το για, για τα περί επιχειρησιακού προγραμματισμού από πλευρά λοιπόν τέτοιου είδου στρατιωτική εμπειρία, αλλά και από πλευρά τη αποστολή σα, η οποία πρόκειται να λάβει τέλο ε, φέτο, γιατί τελικά ε, το χρονοδιάγραμμα καθορίζεται από τη διάρκεια τη κάθε θητεία τη εντολή. Αλλά υπάρχει κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ. Είπατε ότι η Ευρώπη χρειάζεται έναν στρατηγικό βραχείο ισχυρό. Σύμφωνοι σε αυτό η Ευρώπη δεν είναι δυνατόν επαόριστον να γατζώνεται από τον ΝΑΤΟ γιατί θα είναι όλο και πιο σημαντικός ο, ρόλος αυτός της Ευρώπης. Τι εννοείται ακριβώς να λέτε στρατιωτικό βραχείο ισχυρό. χρειάζεται να έχουμε στρατό, εννοείται. Ή εννοείται συντονισμό. Ή εννοείται συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Ή μήπως θα πρέπει να γίνει ένα βήμα παραπάνω. Το οποίο πάει να πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει τις δικές της ένοπλες δυνάμεις. Οπότε, εν τη αυτή περιπτώσει έχουμε το δικό μας στρατό, ποιος θα αποφασίζει την αποστολή σε επιχείρηση αυτού του στρατού. Πώς θα οργανωθεί αυτό. Είδαμε τι έγινε στο Αφγανιστάν. Δεν αρκούν οι επιχειρησιακές μονάδες. Χρειάζεται επιμελητεία, χρειάζεται προγραμματισμός, χρειάζονται υπηρεσίες που θα φροντίσουν για την αποχώρηση των, του προσωπικού. Πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση επίση πόσο θα κοστίσει ένας τέτοιος Ευρωπαϊκός στρατός. Um, General, thank you for being with us and um, I would... Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας κύριε στρατηγέ μου. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα για την CoHQ για το κοινό Στρατηγείο. Θυμόμαστε τι συνέβη με την κυρία Άστον όταν προσπάθησε να προωθήσει αυτή την ιδέα. Προσέκρουσε σε αμετακίνητη αντίθεση από την πλευρά των κρατών μελών. Τι έχει γίνει όμως έκτοτε και ιδιαίτερα οι ιδέες αυτές αποτελούν κατά κάποιο τρόπο τμήμα της ε, αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, αναφέρονται στα πλαίσια της επισκόπησης αυτής που γίνεται και της ενδεχόμενης αναθεώρησης και αν όχι ποιες άλλες ε, οδούς θεωρείτε ότι πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να μπορέσει να καταλήξει σε ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Στρατηγέ μου, έχετε πάρα πολλά ερωτήματα να απαντήσετε. Θα σας έδινα τρεις ώρες για να απαντήσετε, αλλά έχουμε μόνο χαρακαλευτά στην πράξη. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω με τη σειρά που διατυπώθηκαν τα ερωτήματα. Είναι πολλά τα οποία είναι παρόμοια και θα προσπαθήσω να τα ομαδοποιήσω. <clears throat> για το ερώτημα του κυρίου Γκάλερ. Θα ήθελα να υπάρξει και χρηματοδότηση από την ανάπτυξη και την συνεργασία να πληρώνει και για ενέργειες στρατιωτικού χαρακτήρα. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο γίνεται η συζήτηση αυτή και σε εθνικό επίπεδο και πιστεύω ότι πρέπει να σεβαστούμε όλοι τους κανόνες που ισχύουν που προς το παρόν χωρίζουν τους δύο προϋπολογισμούς απόλυτα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν είναι χρήσιμο να υπάρχει συνδυασμό σας πάρουμε την περίπτωση του κέρατος της Αφρικής όπου μπορούν, παραδείγματο χάρη, οι ναυτικέ δυνάμει να εκπαιδεύουν και ακτοφύλακε στι χώρε αυτές. Αλλά δεν μπορούν να αγοράσουν πλοία ακτοφυλακή. Εκεί είναι η γραμμή του προπολογισμού για την ανάπτυξη ασφάλειας σε αυτές τις περιοχές. Επομένως, μπορούν οι στρατιωτικές δυνάμεις να ενισχύουν πολιτικούς τομείς ασφάλειας, αλλά είναι κυρίως στο τομέα της κατάρτισης. Μπορώ να σας δώσω εκατοντάδες παραδείγματα, όπου είναι πράγματι πολύ χρήσιμο να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και αν ζητήσετε ε, να ακούσετε και το Γενικό Διευθυντή για την ε, ανάπτυξη, θα μπορούσε να σας πει και αυτός ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς εξασφάλιση ασφάλειας και εγώ επίσης πιστεύω δεν μπορεί, μπορεί να υπάρξει ασφάλεια χωρίς ανάπτυξη. Νομίζω λοιπόν ότι δεν έχει νόημα να ξοδεύουμε χρήματα για ανάπτυξη όπου δεν μπορούν τα χρήματα αυτά να αποδώσουν αποτέλεσμα ελλείψη ασφάλειας και από τη δική μας πλευρά εμείς δεν έχει νόημα να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια αν δεν ακολουθήσουν πολιτικού χαρακτήρα μέτρα όπως είναι η ανάπτυξη, η ευκυβερνησία, η λειτουργία των αστυνομικών και δικαστικών δυνάμεων κτλ. Και εγώ προσπαθώ να τονίσω ότι θα μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο σε συμμαχίες κατά περίπτωση που έχουν λάβει μέρος σε τέτοιες διαδικασίες. Υπάρχει η υπηρεσιακή ομάδα για το Αφγανιστάν που έκανε ένα θαυμάσιο σχέδιο το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη. Γιατί, Γιατί οι πολιτικοί ε, εμπλεκόμενοι δεν θέλουν να συντονίζονται από τους στρατιωτικούς και οι στρατιωτικοί δεν θέλουν να συντονίζονται από τους πολιτικούς. Επομένως δεν καταλήξαμε πουθενά. Είχαμε την ύπατη εκπρόσωπο, η οποία είχε την εντολή συντονισμού όλων αυτών των εξωτερικών δράσεων. Το κάνει αυτό και εγώ βρίσκομαι στο ίδιο τραπέζι και μπορώ να συντονίζομαι με όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Εκεί είναι το θετικό. Κάποιες φορές είναι τα κράτη-μέλη που οργανώνουν αυτές τις ενέργειες και επομένως ο προπολογισμό που έρχεται από τα κράτη-μέλη και εγώ είμαι στην υπηρεσία των κρατών μελών, κατά συνέπεια και <clears throat> έτσι λειτουργεί το σύστημα. Δεν νομίζω να υπάρξει κάποια τροποποίηση στο άμεσο μέλλον ώστε ο προπολογισμό τη Κομισιόν να χρησιμοποιείται και για στρατιωτικέ δράσει. Για το ερώτημά σα για το συντονισμό με τον ΝΑΤΟ. Εγώ έχω την δυνατότητα να έχω άτυπη συνεργασία με το ΝΑΤΟ και μόνο ε, καταλαβαίνετε γιατί πολιτικού λόγου είναι πιο δύσκολο να έχουμε επίσημη μορφή συντονισμού. Θα ήταν καλύτερα να μην έχουμε τέτοια πολιτικά προβλήματα, αλλά δεν μπορώ εγώ να τα επιλύσω. Εγώ προσπαθώ να πετύχω ό,τι μπορώ στο δικό μου επίπεδο και κάποιοι άλλοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα σε πολιτικό επίπεδο. Όσο λοιπόν εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το πρόβλημα, εγώ τουλάχιστον μπορώ να έχω μια πραγματιστική αντιμετώπιση και γι' αυτό μπορώ να σα εγγυηθώ ότι δεν υπάρχει επικάλυψη με τον ΝΑΤΟ στην ανάπτυξη ικανοτήτων, προσπαθούμε να συνοηθούμε μεταξύ μας σε λογικό επίπεδο και τελικά ό,τι κάνουμε στο ΝΑΤΟ και ό,τι κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αμοιβαία εποφελές. Γιατί, όπως σας είπα, οι στρατιωτικές ικανότητες παραμένουν στα χέρια των κρατών μελών που μπορούν να τις διαθέσουν είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στο ΝΑΤΟ. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο συνδέεται με όλα αυτά. Μήπως είναι λιγάκι ανόητο να γίνεται η ίδια προσπάθεια και από τον ΝΑΤΟ και από εμά για τον, την συνένωση των ικανοτήτων. Μα είναι τα κράτη-μέλη που αποφασίσανε κάτι τέτοιο. Το μόνο που μπορώ να κάνω εγώ είναι να εξηγήσω γιατί μερικές φορές είναι πιο λογικό να επιλέγουμε το ΝΑΤΟ για το γενικό πλαίσιο και ο Γενικός Γραμματέας του ε, ΝΑΤΟ, ο κύριος Γκέιτς, είχε τονίσει ότι δεν είναι θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών το pool and share, η συνένωση των ικανοτήτων. Είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εάν εγώ λοιπόν ήθελα να χρησιμοποιήσω μια ικανότητα που βρίσκεται ήδη στι ΗΠΑ και μπορεί να την υλοποιήσει η Αμερικανική βιομηχανία, εγώ θα προτιμούσα να έχω την υποστήριξη από το ΝΑΤΟ, γιατί τότε θα λειτουργήσει και η Αμερικανική βιομηχανία. Πολύ ωραία. Γιατί για μένα αυτό που έχει σημασία είναι η στρατιωτική ικανότητα. Αν όμω έχετε βιομηχανικές ικανότητες όχι κατά αλλά τροφοδοτικού χαρακτήρα βιομηχανικούς κλάδους που θέλουν και αυτοί να συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας ικανότητας στρατιωτικού χαρακτήρα, τότε εκεί πρέπει να διευκολυνθεί αυτή η, η διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Φορέα. Γιατί ο στόχος αυτού του φορέα είναι να εξασφαλίσει την έρευνα και την ανάπτυξη με την μικρότερη δαπάνη χρημάτων και τον καλύτερο συντονισμό και στην εντολή τους περιλαμβάνεται και το γεγονός ότι θα πρέπει να βοηθήσουν την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, όταν έχει κανείς ισχυρή άμυνα, έχει και ισχυρή βιομηχανία και ισχυρή οικονομία. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό το έργο του Ευρωπαϊκού Φορέα Άμυνας Υπηρεσίας Άμυνας, της EDA κύριε Φανόρντεν. Ένα παράδειγμα μονάχα. Ποιες είναι οι ικανότητες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τον εναέριο ανεφοδιασμό, παραδείγματος χάρη. Εκεί χρειάζεται καλό συντονισμό με τον ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν απλώ να υπάρχει ικανότητα. Θέλει, θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ικανή και να χρησιμοποιεί ευρωπαϊκέ δυνατότητε για αυτόν τον ενάεριο ανεφοδιασμό. Και συγχρόνως έχω ένα άλλο παράδειγμα, όπου νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μια σωστή επιλογή. Εμείς διευκολύνουμε τα κράτη-μέλη να έχουν μια ε, ικανότητα χρησιμοποιώντας τις εναέριες ε, δυνάμεις σχεδίασης που υπάρχουν. Κάθε κράτο μέλο λοιπόν μπορεί να δώσει το δικό του πετραδάκι για να ενισχύσει αυτήν την ικανότητα και παίρνει ένα αντίστοιχο κομμάτι από τι ώρε πτήση. Αλλά μόνο το κράτο μέλο αποφασίζει πώ θα χρησιμοποιήσει αυτέ τι συγκεκριμένε ώρε πτήση. Και όλα τα άλλα κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα δεν μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ώρε πτήση από τα άλλα κράτη-μέλη. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να εξασφαλίσετε μεγαλύτερες εγγυήσεις ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ικανότητες για τις οποίες έχετε καλοπληρώσει. Γιατί πολλές φορές δημιουργείται μία ικανότητα και στη συνέχεια βρίσκεται μονάχα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Αν δημιουργήσετε όμως μία δυνατότητα, μια ικανότητα, ακόμα και αν δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη, αλλά το κάνετε να ανήκει σε ένα οργανισμό ο οποίος λειτουργεί με ομοφωνία, τότε ένα και μόνο κράτος μέλος μπορεί να εμποδίσει αυτή την κινητοποίηση αυτής της ικανότητας. Δαπανάμε λοιπόν εκατομμύρια για μια ικανότητα που να μπορεί να εμποδίζεται από ένα κράτος μέλος. Και η δική μου εμπειρία μου έχει δείξει περιπτώσεις που αυτό να έχει συμβεί. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι μια σοφή αρχή να ακολουθούμε αυτό που είπα προηγουμένως για, την, για τον εναέριο ανεφοδιασμό. Αλλά ένα άλλο παράδειγμα είναι ο στρατιωτικός έλεγχος του εναερίου ε, χώρου. Είχαμε στο παρελθόν τέσσερα κρατημέλη, τώρα έχουμε πέντε κρατημέλη και είναι οργανωμένους με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσει του ΝΑΤΟ, για επιχειρήσει Ευρωπαϊκή Ένωσης για κατά περίπτωση συμμαχίες σε εθνική βάση κτλ. Και κανένα από τα κράτη τα οποία συμμετέχει δεν μπορεί να εμποδίσει τα άλλα κράτη-μέλη από το να χρησιμοποιήσουν αυτή την ικανότητα. Αυτό είναι λοιπόν ο τρόπο με τον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε και αυτή είναι η απάντηση που δίνω στο ερώτημα του αν θέλω να υπάρχει Ευρωπαϊκό στρατό. Είμαι πραγματιστή. Δεν θα με ακούσετε να λέω θέλω Ευρωπαϊκό στρατό γιατί αυτό ξέρω ότι δεν πρόκειται να γίνει για κάθε κράτος μέλος και δεν ξέρω καμία εξαίρεση οι κυβερνήσεις θέλουν να κρατούν την εθνική κυριαρχικότητα σε σχέση με τη χρήση του δικού του στρατού. Και η λέξη κυριαρχικότητας πολλές φορές χρησιμοποιείται καταχρηστικά. Αν δεν θέλει κανείς να συνεργάζεται με τους άλλους <clears throat> λόγω της δικής μας δική σου αντίληψη της κυριαρχικότητας. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι σφάλμα, γιατί η κυριαρχικότητα δεν είναι μονάχα η ελευθερία να αποφασίσει κάνει κάτι. Θα πρέπει ή θα έπρεπε να είναι η ικανότητα δράσης. Αλλιώς είναι περίτη τελείως. Αν είναι κανείς σε ένα νησί και δεν έχει ένα πλοίο και θέλει να φύγει από το νησί, τότε μπορεί να το αποφασίσει, αλλά χρειάζεται και ένα πλεούμενο για να μπορέσει να φύγει από το νησί. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να συνεργάζεται κανείς και με τους άλλους για να έχει τις απαραίτητες ικανότητες. Βαν χωρίς μικρόφωνο. Ο κύριος Μπουτικόφερ, ε, εσείς είστε στο νησί. Είστε στο νησί μόνοι σας. Κύριε, κύριε, λέει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος καλεί τον στρατηγό να πάρετε λόγο. Να συγχαρώ το Ηνωμένο Βασίλειο, να σας κάνω ένα κομπλιμέντο, γιατί κατέφεραν και κατέληξαν σε μια πολύ σοφή σκέψη σε ό,τι αφορά αυτόν τον κοινοεπιμερισμό των εξόδων, γιατί δεν είχε τέτοιες ε, δαπάνες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ήταν δραματική η κατάσταση αν δεν είχαμε τέτοιες δυνατότητε, αλλά σε κάποια φάση, σε κάθε κράτος ε, μέλος, έρχεται κάποια στιγμή που δεν έχει κάνει ε, τα χρήματα ή, εν που η κυβέρνηση αποφασίζει ότι υπάρχουν διαφορετικές ε, προτεραιότητες, ενώ εμείς ως μέλη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε κάποιες ικανότητες και δυνατότητες αν κάποιο κράτος μέλος αποφασίζει να κάνει αυτό το share σε ό,τι αφορά κάποιες τέτοιες δυνατότητες. Και υπήρχε, για παράδειγμα, το παράδειγμα της Γαλλίας, το pooling and sharing, αυτή η κοινός επιμερισμός των ε, εξόδων. Θα υπάρξουν, θεωρώ, καταστάσεις όπου το ΝΑΤΟ καλύτερα θα κάνει να χρησιμοποιήσει δυνατότητες ενός κράτους μέλους. Αλλά θα υπάρξουν και καταστάσεις όπου το ΝΑΤΟ δεν θα μπορέσει να δράσει. Γιατί στην περίπτωση αυτή να μην μπορέσουμε, να μην ε, διασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε από κοινού να προσπαθήσουμε να προσπίσουμε τα κοινά μας συμφέροντα, αν δεν μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας. Αν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας, παρακαλώ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά οι πιο πολλές από τις συγκρούσεις που αντιμετωπίζουμε δεν μπορούν να επιληθούν από ένα κράτος μόνο του. Άρα θα πρέπει να αναπτυχθούν κοινέ δυνατότητες για να εξυπηρετούν ένα κοινό συμφέρον. Διάφορες ερωτήσεις για τον κυβερνοχώρο ακούσαμε και την άμυνα στον κυβερνοχώρο. Μεταξύ των οποίων και μία ερώτηση της κυρίας Κοπά. Να απαντήσω στις ερωτήσεις αυτές ε, από κοινού. Ναι, πρόκειται για σοβαρή απειλή και ναι, μια στρατιωτική απειλή ε, ενέχεται, αλλά ξεπερνά το πλαίσιο της στρατιωτικής ε, απειλής. Και πάλι βλέπω ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη συνεργασία, γιατί πολλοί ανησυχούν σε ό,τι αφορά τον κυβερνοχώρο και ιδιαίτερα από τον τραπεζικό τομέα. Σε ό,τι αφορά βασικά θέματα υποδομών. Εγώ δεν είχα τέτοιο προσωπικό όταν ξεκίνησα, αλλά πολύ είναι περιορισμένο, πολύ περιορισμένη η τεχνογνωσία μεταξύ των ε, ατόμων του προσωπικού μας. Τώρα λοιπόν μπορούμε να συνεργαστούμε και να κάτσουμε να το σκεφτούμε από κοινού για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοιες ε, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Κατά πόσον υπάρχει στρατηγική από πλευρά μου για την αντιμετώπιση των περικοπών. Κοιτάξτε, στρατηγική, μην το πω και στρατηγική. Εγώ θεωρώ ότι εντό του πεδίου των αρμοδιοτήτων μου, αν τα κράτη-μέλη δεν ε, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν κάποιες υποδομέ που χρειαζόμαστε για το κοινό μα συμφέρον, εγώ θα μπορέσω να διοργανώσω μια συνύπαρξη, μια συνεργασία, να προωθήσω πρωτοβουλίες αν ε, είναι σε επίπεδο έργου να τις ε, μεταβιβάσω στην EDA. Αλλά νομίζω ότι για πολλούς ε, λόγους θα καταστεί λειτουργική η όλη υπόθεση μόνο με πολιτική πίεση. Εγώ Έχω συμμετάσχει σε πολλές υπουργικέ συναντήσεις που πολλοί υπουργοί μου λέγαν ότι κοιτάξτε πρέπει να κάνετε αυτό. Αλλά εάν ε, υποβάλω μία πρόταση για κοινή δράση, κάθε κράτος μέλος ξεκινά να προστατεύει τα δικά του συμφέροντα. Άρα τελικά πώς θα γίνει η πρόοδος, πώς θα σημειωθεί η πρόοδος, μόνο αν δεν αναλάβουν αυτοί το δύσκολο κομμάτι. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν πολιτική πίεση σε όλα τα επίπεδα, αλλά και στο στρατιωτικό σκέλος, γιατί αν είναι κανείς, ε, για παράδειγμα, από την αεροπορία, έχει συνειφαστεί με τη μονάδα του. Πώς θα κόψει κανείς δαπάνες από τη δικιά του τη μονάδα για να ενταχθεί σε αυτό το pooling and sharing. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι απαραίτητο. Χρειάζεται λοιπόν πολιτική πίεση από πάνω προς τα κάτω και ακόμα και οι αρχηγοί κυβερνήσεων και κρατών ενδεχομένως να χρειαστεί να ασκήσουν πίεση στους υπουργούς οικονομίας και σε άλλους τομείς για να μπορέσουν να αφήσουν κατά μέρο τα οικονομικά συμφέροντα τα προσωπικά συμφέροντα, τα συναισθηματικά συμφέροντα και το καθεξής. Είναι δύσκολη η διαδικασία αυτή. Κύριε, κύριε Κάμπρη, για την Ευρωπαϊκή Αποστολή στο Μαλί. Νομίζω ότι ήδη απάντησα σε ό,τι αφορά το ερώτημα της ε, κυριαρχίας, σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική ε, επέμβαση, την εισακτική αποστολή στο Μαλί. Δεν είναι στην ατζέντα, αλλά είναι καλό παράδειγμα που καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως έχει δεν μπορεί να κάνει αυτό που έκανε η Γαλλία. Συγχαρητήρια στη Γαλλία, γιατί στο Μαλί θα ήταν καταστροφική η κατάσταση αν δεν, αν δεν είχε ε, επέμβει η Γαλλία. Εμείς είχαμε προγραμματίσει διάφορες δράσεις για να συνδράμουμε στην κατάσταση στο Μαλί, αλλά ήμασταν πολύ απλά υπερβολικά αργοί. Η Γαλλία ήξερε ποιοι κίνδυνοι ενέχονταν και την συγχαίρω για την ταχύτητά της, γιατί η η κατάσταση αυτή θα είχε καταστεί μια ευρωπαϊκή καταστροφή. Είναι τόσο πολλά τα συμφέροντα της Ευρώπης που εμπλέκονται σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία, την ε, το λαθρεμπόριο όπλων. Ξέρετε όλους τους κινδύνους που έχουν να κάνουν με το Σαχέλ, με το Αφγανιστάν και το καθεξήν. Κάτι λοιπόν έπρεπε να γίνει και γι' αυτό λοιπόν ήταν τόσο εύκολο να εξευρεθεί συνένεση προκειμένου να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι μπορεί να κάνει στην παρούσα φάση και αυτό που μπορεί να κάνει είναι να αποστείλει αποστολή για την εκπαίδευση και να δώσει και αρρωγή σε θέματα ε, επιμελητίας. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν υπάρχει σχετικά, σχετικό κονδύλι. Αν το αποφασίσει λοιπόν το Συμβούλιο, θα πρέπει να βρούμε κράτη-μέλη τα οποία θα διαθέσουν και τα, τον σχετικό εξοπλισμό και τα σχετικά μεταφορικά μέσα. Οχτώ χώρες λοιπόν το κάνουν αυτό στην παρούσα φάση και χαίρομαι ιδιαίτερα που το κάνουν. πολλά ερωτήματα μου θέσατε κύριε Φανόρντεν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τις ΕΙΠΑ. Οι ΕΙΠΑ ήταν ξεκάθαρες. Θέλουν και το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη και η ΕΙΠΑ να οργανωθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άλλα συμφέροντα να προασπίσει. Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι είπαν ότι δεν θέλουμε να αποστραφούμε ε, και θέλουμε να παραμείνουμε πιστός εταίρος ως προς την Ευρώπη. Και εμείς το ίδιο πρέπει να κάνουμε προς τις, ε, ως προς τις ΣΥΠΑΣ. Το κάνουμε, αλλά όχι στο βαθμό που θα έπρεπε. Είναι γεγονός ότι αναγκάστηκαν να περικόψουν το σχετικό προϋπολογισμό και να αλλάξουν τις στρατηγικές της προτεραιότητες. Θα είναι λοιπόν όλο ένα και πιο δύσκολο για τη να παρεμβαίνουν και να μας ε, διασώζουν. Και εμείς ως Ευρώπη να περιμένουμε από τον πρόεδρο της Αμερικής να πείθει πάντα τους φορολογούμενούς τους για να μοιραστεί μερίδιο δικής μας κρίσης, για την οποία ε, εμείς φταίμε. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε ένα έθνος, αλλά είμαστε μια ένωση και αποφασίζουμε με βάση κοινέ αξίες. Οι 21 κρατημέλη όντως ε, είναι τα ίδια κράτη-μέλη μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν έχετε κάποια λύση πιο αποτελεσματική, πιο αποδοτική, πολύ ευχαριστώ να την ακούσω και να την ακολουθήσω. Σχόλια εκτό μικροφώνου του κ. Φανόρντεν. Θα με τρομοκρατούσε μια τέτοια λύση, γιατί στην περίπτωση αυτή θα είχαμε κρίσεις που θα μας μπλοκάριζε απόλυτα η προαπέτηση ομοφωνία και δεν θα ήμασταν σε θέση να ακολουθήσουμε τη συνεκτική αυτή προσέγγιση με την οποία προσπαθεί να ακολουθήσει το ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι τα κάλυψα αυτά τη συνεκτική προσέγγιση. Το επόμενο βήμα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε τις φιλοδοξίες μας. Δεν θέλω ε, δεν ζητάω ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την άμυνα, γιατί είναι ουτοπικό. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και νομίζω ότι έτσι απάντησα όλες σας τις ερωτήσεις για τον κύριο Κέλαμ από την Εστονία σας. Ε, συγχαίρω. Συγχαίρω την Εστονία. Νομίζω ότι είσαστε το κατεξοχήν παράδειγμα. Ήταν τεράστια η οικονομική κρίση που μας έπληξε, αλλά εσείς είστε δεσμευμένοι και τηρείτε τις υποσχέσεις σας και επιλύσατε σε μεγάλο βαθμό και την οικονομική την κρίση την ίδια. Επιδείξατε ηγεσία και συχνά χρησιμοποιώ το παράδειγμα της Εστονίας. Συμφωνώ με τον Πολωνό Υπουργό Σικόσκι που έκανε αυτή τη σύγκριση μεταξύ οικονομικής κρίσης και κρίσης ασφάλειας, ε, η οποία ενδεχομένως καραδοκεί. Γι' αυτό ε, και εδώ στο Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια και σε διάφορες άλλες περιστάσεις, γιατί εγώ πρόκειται να αποσυρθώ, αλλά τι θα μείνει μετά από μένα. Είμαστε σε θέση να προσπίσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ για να σας εξηγήσω τι αλλαγές χρειάζονται. Νομίζω ότι κάλυψα τα θέματα για τον κυβερνοχώρο. Ασφαλώς ε, για τη χώρα σας αυτό είναι ιδιαίτερος σημαντικό γιατί είστε και στο ΝΑΤΟ, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση είστε υπεύθυνοι για θέματα κυβερνοασφάλειας και χαίρομαι που μπορούμε να συνεργαστούμε με το ΝΑΤΟ για θέματα Κύριε Σεφοκλέου, ε, σας ευχαριστώ για τα ερωτήματα που μου απευθύνατε. Θα ήθελα να κάνω μία διάκριση σε ό,τι αφορά τη διατύπωση. Υπάρχει πολιτική για την ΚΕΠΑ, αλλά έχει περιορισμούς, τους οποίους τους ξέρουμε. Είναι περιορισμένες οι φιλοδοξίες της. Η κοινή άμυνα είναι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και χρειαζόμαστε το ΝΑΤΟ για την κοινή άμυνα γιατί έχουμε και τις ΙΠΑ αλλά χρειαζόμαστε και τον Καναδά για παράδειγμα. Και ο Καναδάς λοιπόν. Εγώ τι κάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζω ότι δεν αποδυναμώνεται το ΝΑΤΟ και προσπαθώ ό,τι κάνω να ενδυναμώνει το ΝΑΤΟ αντιθέτω. Κυρία Γκόμες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις δικές σας ερωτήσεις. πολύ φοβάμαι σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση. Το δεύτερο ερώτημα που θέσατε. Εξαρτόμαστε από την αλληλεγγύη, από τα κρατημέλη που αποφάσισαν ότι πρόκειται να διοργανώσουν και να χρηματοδοτήσουν μια αποστολή. Αυτό είναι ένα από τα αδύναμα σημεία, ότι ενδεχομένως ε, μια υπουργική συνάντηση να αποφασίσει ότι 27 κράτη-μέλη θα συνδράμουν για την διοργάνωση μιας αποστολής και όταν ζητάω τελικά το σχετικό εξοπλισμό, όλοι κοιτούν το ταβάνι. Πώς θα βελτιωθεί αυτό? Όλοι θα πρέπει να αποφασίσουν ότι όταν λαμβάνετε μια κοινή απόφαση όλοι θα συμμετέχουν έστω οικονομικά. Το ΝΑΤΟ παρεπιπτόντως έχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Και εκεί πρέπει να βελτιωθεί η κοινή χρηματοδότηση για τις κοινέ αποστολές. Γιατί πολλές φορές παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο, όλοι περιμένουν από τους άλλους να, να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Δεν γίνεται όμως έτσι. και συχνά βλέπω πολλούς ε, συναδέλφους σε όλα τα επίπεδα που δεν κατανοούν ακόμα γιατί χρειάζεται πολιτικό σκέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε Είναι 200 μόνο οι στρατιωτικοί, ξέρετε, στην... στο προσωπικό μου. Μόνο. Είμαστε 7.500 και δεν περιλαμβάνονται καν αυτοί του IMS, του ΝΑΤΟ. Αυτό κάνει τη διαφορά. Και πολλοί στρατιωτικοί έχουν πολύ πιο πολλές πολύ πιο πολλή εμπειρία στο ΝΑΤΟ παρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ήταν η πρώτη θέση που είχα, η πρώτη λειτουργία που είχα στη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε κοινή διοργάνωση με το ΝΑΤΟ. για τον κύριο Κάμπελ. Α, μάλιστα. Α, νομίζω σας εκάλυψα προηγουμένως. Για τον Όρθουρ ρωτήσατε. That NATO uh, and other people... Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το που λένε για τον ΝΑΤΟ. Ε, που λένε ότι υπάρχει κάποιο είδου επικάλυψη. Ενώ την άλλη μεριά υπάρχει απόφαση συντονισμού σε επίπεδο Γενικών Γραμματείων μεταξύ ημών και εκείνων και μεταξύ του Προέδρου από την άλλη μεριά της Στατικής Επιτροπής και με τις πολιτείες ότι θεωρούν ότι είμαστε η ομολογή τους και μας αναθέτουν να κάνουμε κάποια πράγματα. Και γιατί αυτό, γιατί το πρόβλημα δεν βρίσκεται στις δυνάμεις κατά θάλασσα, στο ναυτικό. Το, προ... το πρόβλημα είναι σε περιπτώσεις όπως η Σομαλία. Και αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την πειρατεία, ε, τότε χρειαζόμαστε πολύ να εμπλακούν και από κοινού να λύσουν το πρόβλημα. Η απάντηση ποια ήταν ότι προτιμούσαν αυτό να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως το ενδιαφέρον που τώρα μου προέγυψε είναι ότι ε, βεβαίως αναγνωρίζεται το ότι είναι χρήσιμο να συνεχίσει το ΝΑΤΟ να χρησιμοποιεί τις ομάδες, τις δυνάμεις, τις, κλασικέ που είχε, θα πρέπει αυτό να, να, συνεχίζουν, να, συνεχίζουν το κάνουν και αυτό και να συγχρησιμοποιούν τις μονάδες αν ΕΡΕΦ για τέτοιου είδου πολέμου. Άρα δεν πρόκειται εδώ για επικάλυψη ενεργειών. Πρόκειται για εξάρτηση των δυνατοτήτων. Αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε πιο άρτια εντολή. Διότι μπορούμε να προβούμε σε συνεννοήσει με τις γειτονιάζουσε χώρες που μπορούν εκείνοι να παραπέμπουν στη δικαιοσύνη του πειρατές που εμείς εχμαλωτίζουμε. Άρα χρειάζεται κάποιο είδου πιο στεγανό νομικό πλαίσιο ως προς το ΝΑΤΟ γιατί έχουμε διπλωματικές δυνατότητες, αναπτυξιακές και... Εντάξει, δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε για τους πρόεδρους, αλλά δεν μπορούσε να γίνει άλλο τους διαδοχή και έτσι βελτιώνουμε τους φορείς όπως η ΣΥΤΡΑ. Γιατί επομένως να μην έχουμε καλύτερη εντολή και επίσης να μπορούμε έτσι να τους επιτεθούμε στο, των πειρατών δηλαδή και κατά ξηρά. Η εντολή επομένω το εξηγεί. Και είναι αστείο το ότι ενώ αναλαμβάνουμε πάρα πολύ ευθύνε αποστολές κατά θάλασσα, για από την άλλη μεριά έχουμε αυτόν τον στόχο που είναι παιχνιδάκι και δεν μας επιτρέπει η εντολή μας να τον ακουμπήσουμε. Άρα το ΝΑΤΟ θα πρέπει να μας βοηθήσει να έχουμε την άρτια εντολή. Γιατί υπήρχαν μια σωρό χώρε που αναρωτιόνται γιατί να μην μπορούμε να αναλάβουμε κατά ξηράν δράσει στην Σομαλία ούτω ώστε να απειλήσουμε την σύγκρουση. Η απάντηση είναι ε, αυτό που κάθεται δίπλα σε μένα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αυτό μπορεί να το κάνει. Και είπε στο Συμβούλιο ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ. Αν μπορούσατε ω Ένωση να λάβετε αυτέ τι ενέργειε, διότι η πειρατεία αποτελεί την ταφόμπλακα στην ανάπτυξη. Είναι κακό για την οικονομία. Είναι κάτι κακό και για τον τουρισμό. Χρειάζεται επομένω καλύτερο συντονισμό και όπως και εσείς συνεπέρανα το ίδιο. Με καλύτερο συντονισμό θα είχαμε καλύτερο σύστημα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ε, of the military action. Όσον αφορά τις στρατηγικές επιχειρήσεις, καθαρά. Πρόκειται για επιτυχία, τακτική, στρατιωτική φυσικό ότι καταφέραμε να τους βυθίσουμε, να τους καταστρέψουμε πλοία τέλο πάντων και τους κινητήρες μαζί, τις μηχανές. Ήταν στρατηγική, όχι μόνο στρατιωτική επιτυχία, γιατί επίσης μέσω του συντονισμού διπλωματικής οδού κλπ. μέσω της καλής συνεργασίας με τις τοπικές αρχές, δημοσία. Έγινε γνωστό ότι στηρίζονται οι ενέργειές μας διότι θα πρέπει να απαλλαγούμε από την πειρατεία. Έτσι αλλάζει η κατάσταση στη Σομαλία και ήταν μια πολύ σημαντική αλλαγή η οποία είχε στρατηγική σημασία. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει σε άλλο οργανωτικό πλαίσιο αυτό. Και όπως ελέγχθη προηγουμένως, ε, εργάζομαι στην υπηρεσία των κρατών αλλά είμαστε όλοι μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπηρετούμε όλοι τις γενικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προσβλέπω στο να εμπλακούν οι δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα από τις αρχές αυτές και θα ήταν και ε, επικίνδυνο τη στιγμή που οι αποφάσεις λαμβάνονται κατ' ομοφωνία. Θα μπορούμε να κινητοποιήσουμε δυνάμεις που να μην μπορούμε μετά να τις χρησιμοποιήσουμε. Στον κύριο Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Όπως ε, είπα προηγουμένως, δεν προσβλέπω σε ένοπλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλώς να υπάρχουν επαρκείς ικανότητες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο εκπονούμε και φέρουμε σε πέρα τις επιχειρήσεις μας. Αυτό που κάνουμε είναι πολύ πιο περιορισμένο από αυτά που κάνουμε στο ΝΑΤΟ το να το ήδη κάνει αυτά τα πράγματα και γνωρίζει πώς να τα κάνει, εμεί χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες με τον ίδιο τρόπο που τις χρησιμοποιεί. Παίρνουμε και εμείς τις πληροφορίες από τα κράτη-μέλη όπως και το ΝΑΤΟ. Το κράτος μέλος δίνει τις πληροφορίες στο ΝΑΤΟ, τις δίνει σε μένα, συν... τις αξιολογούμε στα πλαίσια των σενάριων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΝΑΤΟ μέσα στα πλαίσια των σενάριων του ΝΑΤΟ και νομίζω ότι δεν πρέπει να κινητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη προς την κατεύθυνση ενός ευρωπαϊκού στρατού, λαμβανομένης υπόψη της μορφής λήψης αποφάσεων αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ πρόημο λοιπόν, είναι πολύ πρόωρο για να σκεφτούμε μια τέτοια επιλογή. Δεν θα λάβει χώρα στη δική μου ζωή τουλάχιστον. Και το τελευταίο ερώτημα. Ναι, ναι, ναι, το, το θυμήθηκα τώρα. η ύπατη εκπρόσωπος δεν ήθελε να υπάρξει ένα μόνιμο αρχηγείο στρατιωτικών δυνάμεων. Δεν το επεδίωξε και αυτή ήταν και η δική μου συμβουλή και η συμβουλή όλων των άλλων δομών που την αρρωγούσαν. Το μόνο πράγμα που ήθελε και ήταν απόλυτα λογικό είναι όπως έχουμε στρατιωτικούς, πολιτικούς σχεδιαστές για την, ε, σε αστυνομικέ δυνάμει και για την τήρηση της τάξης και όλοι θέλουν να εξασφαλίσουν να είναι συνολική η σχεδιασή τους και το ίδιο κάνουμε και για την ανθρωπιστική και ανακοφιστική βοήθεια γιατί να μην έχω 20 σχεδιαστές για τις μη ε, εκτελεστικού χαρακτήρα ενέργειες. Όσοι λένε ότι αυτό είναι επικάλυψη με τον ΝΑΤΟ, εντάξει, μα και εγώ έχω σχεδιαστέ. Το ΝΑΤΟ έχει πολύ περισσότερους βέβαια. Εγώ ζητώ απλώς να έχω ένα μικρό περιορισμένο αριθμό σχεδιαστών, ώστε για τις στρατιωτικές αυτές αποστολές που θα ήταν γελίο να κινητοποιήσουμε ένα στρατηγείο με 250 άτομα, όπου μπορεί να γίνει αυτό με 15-20 άτομα και χρησιμοποιώντας τους σχεδιαστές πολιτικής Αλλά επειδή γνωρίζω και τη μία πτυχή και τη στρατιωτική πτυχή και επειδή κάνω επιχειρησιακή σχεδίαση το μεγαλύτερο τμήμα της ζωής μου, αν έχω 20 μονάχα γενικούς επιτελικούς και μπορώ να και πρέπει να δώσω υποστήριξη σε μια εκπαιδευτική ενέργεια στο Μαλί, στην Σομαλία ή όπου αλλού χρειαστεί. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτούς τους σχεδιαστές ως ένα βασικό πυρήνα, οι οποίοι μπορούν να συντονίσουν τα πάντα, τις υποδομές, τις ε, υγειονομικές υπηρεσίες, να αντιμετωπίσουν τα θέματα αποφυγής των συγκρούσεων κτλ. Μπορούν να το κάνουν αυτό. Νομίζω ότι αυτό μας δίνει το χαμηλότερο κόστος Αν μπορώ να χρησιμοποιήσω λοιπόν ένα κέντρο το οποίο είναι ενεργό μόνο για τη Βόρεια Αφρική, να το χρησιμοποιήσω και για άλλε κρίσει οι οποίε θα έχουν στη συνέχεια, αυτό είναι τζάμπα. Απλώ χρειάζεται η πολιτική συμφωνία που θα μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω αυτέ τι ε, ικανότητε και θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν αυτοί οι οποίοι ακόμα τροχοπεδούν αυτές τις όσο απλές αποφάσεις το επανεξετάσουν. Σίγουρα μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο που εκμεταλλευόμαστε τις ικανότητες που έχουμε ήδη τώρα. Αν προτού πάω στη σύνταξη έχω αυτή την υποστήριξη από εσά, θα είναι θαυμάσιο. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε, στρατηγέ μου, για τα σχόλιά σας, για τις απαντήσεις σας. Πάντα πάρα πολύ σαφή αυτά που μας είπατε και πολύ σημαντικά. Ίσως μπορούμε να ξαναβρεθούμε και σε μια άλλη χρονική στιγμή, αν όχι με την τωρινή σας ιδιότητα, πάντα μπορούμε να ξαναβρεθούμε σε συνδιασκέψεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν και εξ ονόματος όλων των μελών της υποεπιτροπής μας για τη συνεργασία σας μαζί μας. Ladies uh, Κυρίες και κύριοι, προχωρούμε τώρα. Περνάμε από την ξηρά στη θάλασσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει κάποιες ενέργειες όπως η επιχείρηση Αταλάντα και η δεύτερη αποστολή Νέστορ. Είναι ακόμα πιο σημαντική. Αυτές είναι οι ναυτικές μας δραστηριότητες. Και ερχόμαστε στην έκθεση της κυρίας Γκόμες από την Σοσιαλιστική Ομάδα για την θαλάσσια διάσταση της, της ΚΕΠΑ. Και επειδή έχουμε καθυστερήσει λιγάκι, δίνω ακαριέα το λόγο στην κυρία Γκόμες. Σας ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για πρώτη φορά προσπαθούν να αναπτύξουν μια τέτοια στρατηγική για την ασφάλεια της θάλασσας. Από ό,τι μου λένε, πριν το θεωρώ έχουμε ένα έγγραφο εργασία, οπότε και η επίσημη πρόταση πρόκειται να υποβληθεί στο Συμβούλιο ε, Αμήνη τον Δεκέμβριο. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση για μα είναι μια ευκαιρία, ούτω ώστε να μπορούμε να επηρεάσουμε τη ζήμωση, την προβληματική, να ακουστεί η φωνή του Κοινοβουλίου και ότι λαμβάνονται υπόψη αυτά που πρεσβεύουμε. Αυτή η στρατηγική χρειάζεται να άρει το κενό το οποίο υπάρχει από την ολοκληρωμένη πολιτική για τη θάλασσα που εγκρίθηκε το 2007 και που ουσιαστικά δεν φύγει την ε, πτυχή άμυνας και ασφάλειας. Θα πρέπει να βασιστεί σε εκείνη την θαλάσσια πολιτική, αλλά επίσης, που πολύ σημαντικό, θα πρέπει να έχει ως θεμέλιο και την πολιτική ασφάλειας. Στην έκθεση αυτή, για αυτό το λόγο, Προσπαθώ να τονίσω το πόσο χρειάζεται μια τέτοια στρατηγική για την ασφάλεια στη θάλασσα και εκεί να την υπόψη τα διακυβεύματα, οι κίνδυνοι, οι απειλές, οι ανάγκες αλλά και οι ευκαιρίες που έχει να αντιμετωπίσει κατά θάλασσα η Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια να φύγεται και το θέμα της προστασίας των Ευρωπαίων. Όμως, επιτύχοντας το μας θα πρέπει να κινητοποιήσουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα θεσμικά όργανα, παράγοντες, μέσα, εργαλεία και πολιτικής και στρατιωτικής φύσεως. Και όμως και σε άλλες πολιτικές μας που έχουμε συζητήσει και προκειμένου έχουμε τα μέσα αυτά τα οποία χρειάζονται, τόσο ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση, το οποίο αφορά και την ασφάλεια και την άμυνα, αλλά η μεγάλη πρόκληση είναι πώς ε, θα αποδώσουν αυτά τα μέσα για αυτόν τον σκοπό μας, πώς θα αποφύγουμε τις επικαλύψεις σε κόστος, σε, σε πόρους, έχοντας την υπόψη επομένως και τη συγκυρία της κρίσης, ώστε να μπορέσουμε το pooling και sharing να το υλοποιήσουμε. Ίσως να περισσώσουμε θέσεις εργασίας, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας που έχουν σχέση με τους κλάδους που κατασκευάζουν το υλικό, τον εξοπλισμό που χρειαζόμαστε. Τι σημαίνει όλα αυτά στην πράξη, τι χρειαζόμαστε. Έχω γράψει στην εκθεσή μου ότι θα πρέπει πρώτα πρώτα να επισημάνουμε ποια είναι τα μέσα, ποιε είναι οι δυνατότητε που θα πρέπει να έχουμε, όταν συνειδητοποιήσουμε τις τι απειλέ σε σχέση με την, την ασφάλεια κατά θάλασσα. Χρειάζονται ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, χρειάζεται εποπτεία, έλεγχο, επαγρύπνηση σε σχέση με την ευρωπαϊκή ακτοφυλακή αναζήτηση, διάσωση ε, και ένωση. Και θα πρέπει κατά θάλασσα να συμπληρωθεί από πολιτικά μέσα η πά, εμπάργκο, ανάλυση παραστάσεων, απεικονίσεων. Ας πούμε, είδαμε τι έγινε στη Σομαλία. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που καταφέραμε όπως επιστώθηκε και έτσι μπορούσαμε πάρα πολλά από αυτά που σας είπα να τα καλύψουμε. Όμω θα πρέπει να είμαστε ε, έτοιμοι να μπορέσουμε να κάνουμε τα ίδια και αλλού. Και αλλού όπου αντιμετωπίζουμε κάποιε προκλήσει και απειλέ. Να μπορέσουμε επομένω κάτι να κάνουμε επιτέλου για τόσα διαδραματίζοντα στο Σαχέλ στην Βόρεια Αφρική. Βλέπουμε ότι όσα γίνονται εκεί είναι πάρα πολύ βασικά και εκτό από και κατά θάλασσα ενδεχομένω έχουμε αντιμετωπίσει αυτές τις ε, προκλήσεις. Είδαμε το πώ ε, στο Σαχέλ ε, λειτουργούν οι τρομοκράτε σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Εκεί έχουν δίκτυα και ήδη, ήδη δρούν και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ακόμα και υποβρύχια έχουν. Ξέρετε, οι έμποροι των ναρκωτικών τα χρησιμοποιούν τα υποβρύχια για να συνδέσουν Νότια Αμερική με Δυτική Αφρική. Με στόχο δε την Ευρώπη. Μιλούμε τώρα για ιδιώτες, για φυσικά πρόσωπα, για κράτη που έχουν υποβρύχια. Επίσης. Θα πρέπει η διπλή χρήση και τεχνολογία να αναπτυχθεί, να προχωρήσει και έτσι να αντιμετωπίσουμε την κρίση ως αρνητικό παράγοντα σε επίπεδο εθνικού προπολογισμού. Επίσης θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη που περιβρέχονται από θάλασσα να έχουν ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες οδηγούν σε υλοποίηση του pooling and sharing, πρόκειται για πρωτοβουλίες με καλή σχέση αποτελέσματος Χρειάζομαστε ακόμα καλύτερη συνάρθρωση και συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Πήγα στην Άμσα, ξέρετε, την υπηρεσία που ασχολείται με την ασφάλεια κατά θάλασσα που έχει έδρα την Λισαβόνα. Φανταστικό είναι το έργο το οποίο εκεί επιτελούν. Και διαπίστω ότι συνεργάζονται με την Ατλάντα με την ΕΣΟ, με την επιχείρηση Αταλάντη. Και όλα αυτά άτυπα. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά για την επιτυχία του Αταλάντη. Μα πώς γίνονται και όλα αυτά γίνονται ενώ δεν προβλέπονται θεσμικά. Γίνονται διότι για να εξυπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο σκοπό έχουν επιστρατευθεί και πολίτε και στρατιωτικοί. Προσπάθησα να τονίσω στο κείμενό μου ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποιες είναι οι προκλήσεις. Ε, αλλά εδώ πέρα υπάρχουν και οικονομικές ευκαιρίες. Εδώ ξανοίγονται εμπορικές ευκαιρίες. Να, όσον αφορά την διόρυγα του Παναμά. Δεν αλλά όμως θα ξανοίξει του χρόνου. Του χρόνου. Και έτσι θα έχουμε διευκόλυνση της επικοινωνίας των δύο ωκεανών. Στην Αρκτική επίσης ξέρουμε τι προβλήματα υπάρχουν και γνωρίζουμε όμως ότι περισσότερη εμπορική ροή σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη ασφάλεια που να προστατεύει τις εμπορικές ροές. Και έτσι θα υπάρχει βέβαια και επίπτωση βία το περιβάλλον. Και έτσι θα απαιτείται περισσότερη επαγρύπνηση. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα τομέα που μπορούμε πραγματικά να επηρεάσουμε τα όσα επιτελεί η Κομισιόν στην υπηρεσία εξωτερική δράση. Μπορούμε να έχουμε όραμα, μπορούμε να έχουμε, λέγω στην έκθεση, αισιοδοξία, φιλοδοξία. Πρόκειται για για την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Και Πρώτη για άμυνα και ασφάλεια εδώ. Ακόμα και για να αντιμετωπίσουμε την απειλή από την αλλαγή του κλίματος. Βεβαίως, μια που εγώ δεν είμαι ειδική, θα βρεθούν πιο ειδικοί από μένα. Και γι' αυτό σας λέω. Είμαι βέβαιη ότι θα βοηθήσουν διάφοροι συνάδελφοι αλλά και διάφοροι εξειδικευμένοι φορείς. Οπότε και με τη βάση του κειμένου που έφτιαξα θα έχουμε μια έκθεση πιο φιλόδοξη, πιο στοχευμένη. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιδράσουμε εις ό,τι πάνε να αποφασίσουν στο επόμενο Συμβούλιο Άμυνα τα κράτη. μέλη. Ευχαριστώ κύριε Αγκόμε. Ο πρόεδρο του ο κύριο Ντανζόνιος και ο δισηγητή από το ΕΛΚΑ, επειδή είναι απόν, θα ήθελα να ζητήσω από τον Μάικελ Γκάλαρ, τον συντονιστή, να πει δύο-τρία λόγια για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο Αρνό λείπει, αλλά τα σχόλια του είναι παρόντα. Μπορώ να σας τα μεταφέρω εξ ονόματός του. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συγχαρεί, Άννα, για την πλήρη αυτή έκθεση, την εμπεριστατωμένη αυτή έκθεση. Εξηγεί η έκθεση γιατί πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ενεργή στη θαλάσσια πολιτική, ποια είναι τα συμφέροντα τα οποία μπορεί να υποστηρίξει, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των ωκεανών και των παράκτιων περιοχών. Η έκθεση αυτή επίσης ορθά εισάγει τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως εμπλεκόμενος στα διεθνή θέματα της θαλάσσιας ε, ασφάλειας, είτε είναι οργανωμένα δίκτυα, εγκληματικά, είτε είναι πειρατές, οι γεωγραφικές περιοχές πρέπει να είναι ε, ενεργοί στην ε, ε Βαλτική, στην ε, Μαύρη Θάλασσα, στη Μεσόγειο, στον κόλπο της Γουινέας, στον κόλπο του Άδεν, στην Αρκτική κτλ. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση σε όλες τις προκλήσεις για την ε, θαλάσσια ασφάλεια και επίσης χάρη στην έγκριση αυτής της πολιτικής υπάρχει η θέληση δημιουργίας εταιρικών σχέσεων με άλλους εταίρους. Ο στόχος έκθεση να προωθήσει τη δημιουργία ικανότητα στον θαλάσσιο χώρο, ιδίως ό,τι αφορά την επιτήρηση, τις περιπολίες και την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου το οποίο θα μπορέσει να συναρθρώσει καλύτερα τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήδη υφίστανται και να συντονίσει καλύτερα την ναυτική και θαλάσσια πολιτική των κρατών μελών. Και υποστηρίζει επίσης η έκθεση πρωτοβουλίες όπως η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής. Ο κ. Νταουζάν όμως θα ήθελε να αναφέρει και ορισμένα σημεία τα οποία κατά την άποψή του θα ενίσχυαν αυτή την έκθεση. Πιστεύει ότι η έκθεση δεν εστιάζει επαρκώς στον κύριο τίτλο της έκθεσης που είναι η ΚΕΠΑ, γιατί ο τίτλος της έκθεσης είναι η θαλάσσια διάσταση της ΚΕΠΑ, ενώ η έκθεση κυρίως ασχολείται με την στρατηγική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη θάλασσα. Αφορά βέβαια θέματα που έχουν την ΚΕΠΑ, θέματα ανάπτυξης, θέματα αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων, κοινωνική και ε, ε, άλλε μορφέ ανάπτυξη. Κάποια από αυτά τα θέματα είναι τμήμα τη συνολική προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια και είναι σημαντικό να αναφερθούν, αλλά ο κ. Ντανζόν πιστεύει ότι αυτά είναι κάπως σε βάρος της ίδιας της ΚΕΠΑ που πρέπει να είναι το κεντρικό θέμα. Αναφέρεται στην παράγραφο 11 λέει ότι επιτέλους αναφέρεται η ΚΕΠΑ στην παράγραφο αυτή. Η έκθεση λοιπόν θα μπορούσε να δώσει περισσότερη έμφαση στην ε, επιχείρηση Αταλάντα, την επιχείρηση στο κέρας της Αφρικής που ήταν μια ιδιαίτερα επιτυχής έκφραση της θαλάσσιας διάσταση της ΚΕΠΑ και μπορεί να αποτελέσει και θετικό υπόδειγμα για μελλοντικές ενέργειες. Και τέλος, λέει ο κ. Δανζόν, θα πρέπει να εστιάσει και περαιτέρω η έκθεση αυτή στις εταιρικέ σχέσεις οι οποίες θα μπορούν να γίνουν σε διάφορες περιοχές όπως ο Νότιος Ειρηνικός, όπου είναι δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει τις δυνάμεις της, αλλά που μπορούμε να βρούμε εταίρους. Σας ευχαριστώ. Thank you, Arnold. Thank you. Σας ευχαριστώ, Άννα, σας ευχαριστούμε, Μάικλ, κυρία Νικολάη από την Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν θυμάστε, το 2007 ξεκινήσαμε να σχολιάζουμε τις ελλείψεις της θαλάσσιας πολιτικής και τώρα μιλάμε σε ό,τι αφορά τις ανάγκες ε, του σχεδίου. Έξι χρόνια έχουν μεσολαβήσει, πολλοί χρόνος αλλά πραγματικά χρειάζεται η τομεακή αυτή η τομεακή προσέγγιση σε ό,τι αφορά την θαλάσσια ασφάλεια και άμυνα. Καταδεικνύετε στην έκθεσή σας γιατί χρειάζεται αυτή η στρατηγική. Αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για να ορίσουμε από κοινού το πώς θα καταρτιστεί αυτή η στρατηγική. υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και συμβολής του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της ε, θαλάσσιας διάστασης της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Δεύτερο θέμα είναι γεγονός ότι πολλά κράτη-μέλη εξαρτώνται από τις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά ο μοναδικός τρόπος είναι να δημιουργήσουμε εταιρικές σχέσεις σε όλο το τομέα των ε, συμφερόντων των κρατών μελών. Τρίτον, ε, τομείς έντασης σε ό,τι αφορά κράτη και σε ό,τι αφορά τον ε, αρκτικό χώρο. Καλωσορίζω την σχετική σας προσέγγιση. Θα μπορούσαμε και στο σημείο αυτό να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τις σχετικές διαφορές. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και να και θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες προσεγγίσεις, συγκεκριμένα σχέδια σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη μας και εκείνη μας δράση. Τελευταίο θέμα για το πώς θα συνενώσουμε τις δυνάμεις μας για να πετύχουμε τα όσα θέλουμε να πετύχουμε στην θαλάσσια πολιτική. Και αυτό αφορά τις ε, χώρες που έχουν πρόσβαση στη θάλασσα και τις περίκλειστες χώρες. Θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση τελικά θα αφορά όλες τις χώρες, ακόμα και αυτές που δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, γιατί όλοι μας θέλουμε να προασπίσουμε την οικονομική μας ασφάλεια και η Αταλάντη μας δείχνει ότι ακόμα και ένα περιστατικό στο κέρας της Αφρικής μακριά από μας επηρεάζει τις χώρες μας. Θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες, αλλά εν γέννη υποστηρίζουμε την έκθεση, συμφωνούμε με πολλά στοιχεία που περιλαμβάνει και νομίζω ότι αν συνεργαστούμε θα είναι πολύ επιτυχής η έκθεση αυτή και πολύ χρήσιμη. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, εξ ονόματος των Πρασίνων, ο κύριος Μπεντικόφερ που φοράει και πράσινη γραβάτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γενικά, δεν υποστηρίζουμε τη φιλοδοξία που προασπίζει αυτή η έκθεση και θα ήθελα να υπογραμμίσω εξ αρχής δύο σχόλια τα οποία διάβασε ο κύριος Γκάλερ τα σχόλια του κύριου Τάντζον, του Πρόεδρου. Αυτό που μου λείπει εδώ είναι κατά πρώτον μία επικέντρωση στην ΚΕΠΑ και κατά δεύτερον μία επικέντρωση, επικέντρωση σε στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις. Να σας εξηγήσω κάποια από τα κριτικά μου αυτά σχόλια. Τα επικριτικά μου αυτά σχόλια. Στο Α η έκθεση μιλάει για την ακτογραμμή της Ευρώπης και αυτό ασφαλώς συνδέεται με την πρόταση του 44 για την δημιουργία Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Δεν θεωρώ ότι αυτό το προδιαγράφει η συνθήκη και δεν, το, δεν είναι στο πεδίο αρμοδιότητας της ΚΕΠΑ. Μιλάμε για το εξωτερικό εμπόριο. Να σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με την συνθήκη η ΚΕΠΑ θα πρέπει να επικεντρώνεται στα καθήκοντα όπως η ειρήνευση, η επιβολή της ειρηνής και η διάσωση. Δεν θεωρώ, δεν υπάρχει μάλλον σχετικός ορισμός στην συνθήκη που θα μας επέτρεπε να προωθήσουμε τους στόχους που περιλαμβάνονται στο Β, στο σημείο Β. Και αυτό επανέρχεται και στην παράγραφο 1. Η ΚΕΠΑ δεν αφορά μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία του ευρωπαϊκού εμπορίου. Στην παράγραφο 2, Άννα, προτείνεις η Ένωση να επιτελέσει το ρόλο της ως πάροχο παγκόσμιας ασφάλειας και να παρέχει οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά και το καθεξής επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο. Το συγκείμενο, το πλαίσιο δείχνει ότι θέλετε αυτό να το κάνουμε χρησιμοποιώντας στρατιωτικά μέσα. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αρμοδιότητα καθήκον στα πλαίσια της ΚΕΠΑ. Δεν είμαι καθόλου βεβαίως κατά πόσον μάλιστα αυτό θα βελτίωνε την ασφάλεια της Ένωσης και των πολιτών. Δεν υπάρχει κοινή πολιτική για την άμυνα. Αυτό είναι γεγονό και ούτε θα έπρεπε, θεωρώ, αναγκαστικά να αποτελεί στόχο μας. Ίσως θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να συζητάμε θέματα σχέσεως ε, ΚΕΠΑ και ΝΑΤΟ. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα πρέπει να ορίσουμε την ΚΕΠΑ. Ακόμα και σε μελλοντικό επίπεδο ως κάτι που θα υποκαταστήσει την κοινή αυτή στρατηγική άμυνας. Θα προτιμούσα να κοιτάτε θέματα εταιρικής σχέσεως, όχι μόνο με τον ΝΑΤΟ, αλλά και με τον ΝΑΤΟ. Κάποια συγκεκριμένα θέματα σε ό,τι αφορά τον ευξηνοπόντο, παράγραφος 17 κατά πόσον θα ήταν ε, δυνατόν πάλι υπό την κεφαλίδα της εταιρική σχέσης να κοιτάξουμε θέματα κοινή στρατηγικής ε, στον εύξηνο πόντο σε ό,τι αφορά την παράγραφο 22 ίσως χρήσιμο θα ήταν να αναφερθούμε στο ρόλο που διαδραμάτισαν στο πλαίσιο αυτό οι ευρωπαϊκές εταιρείες στην παράγραφο 26 δεν είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τον στόχο της δημιουργίας ε, ναυτικής βάσης στο πράσινο ακροτήρι. Στην παράγραφο 30. η συνεκτική προσέγγιση, αυτή η συνολική προσέγγιση και η υποστήριξη της αρχής αυτής που θεωρείται ότι είναι κάτι το δεδομένο στο κέρας της Αφρικής, εγώ δεν τη βλέπω πουθενά παραγράφος 31 και 32. Και οι δύο μιλούν για την Αρκτική. Και πάλι όμως δεν βλέπω πουθενά το θέμα της συνεργασίας με το Συμβούλιο της Αρκτικής. Δεν θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε, λες, και δεν υπάρχει κανένα απόλυτο σώμα με το οποίο μπορούμε και πρέπει να συνεργαστούμε. Παράγραφος 33. Καταρχάς, να σας πω ότι Δεν μιλάμε μόνο για την ε, θάλασσα της Νότιας Κίνας. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να μιλάμε για τη θάλασσα της Νότιας Κίνας, γιατί υπάρχουν και άλλες ε, χώρες στην περιοχή που προετοιμάζουν άλλα νόματα και ίσως θα πρέπει να την αποκαλούμε με τρόπο που να μην ε, δείχνει προκατάληψη προς ένας από τις δύο, προς, μία από τις χώρες αυτές. Και πάλι θα πρέπει να συνεργαστούμε με τη Σιγκαπούρη σε ό,τι αφορά θέματα θαλάσσιας επιτήρησης για ειρηνικού σκοπούς. Και αυτό θα μπορούσαμε να το αναφέρουμε εδώ πέρα. Αλλά αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 34, αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 34 με σοκάρει. Αναφέρεται ότι καλεί την ύπατη εκπρόσωπο αντιπρόεδρο κατεπηγόντως να εντοπίσει τα μέσα και τις δυνατότητες ιδιαίτερα τις θαλάσσιες δυνατότητες που ενδεχομένως θα χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναπτύξει στην περιοχή, για να προασπίσει τα συμφέροντά της και, και να προλάβει συγκρούσεις και ούτω καθεξής. Δεν μιλάμε για θέματα πραγματικότητας. Δεν νομίζω ότι θα ήταν έξυπνο, ακόμα και αν είχαμε σχετικό στόλο να θέσουμε τέτοια θέματα σε ό,τι αφορά τον ελληνικό. Στην 37. Δεν μετανιώνω εγώ προσωπικά που έγιναν περικοπές στον προπολογισμό για την άμυνα. Αυτό που με λυπεί είναι που δεν χρησιμοποιούμε τις περικοπές αυτές που έγιναν για να κινηθούμε πιο φιλόδοξα προς την κατεύθυνση του pooling and sharing και ελπίζω να μπορέσουμε να προσθέσουμε κάποια έκφραση που θα έχει να κάνει με την ανάγκη ιδιωτική ασφάλισης στον τομέα των θαλάσσιων. Παράγραφος 31. Δεν συμφωνώ με την αναφορά ότι η βιομηχανία της άμυνας ε, έχει να κάνει με τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν θεωρώ ότι αυτό περιγράφει καταλήλω την κατάσταση στη Γερμανία. Θεωρώ ότι η έκθεση αυτή λοιπόν είναι εξαιρετικά υπερφιλόδοξη πέρα του δέοντος. Περνά πολύ πέρα από τον αρχικό της στόχο, ο οποίος είναι να εξεταστεί η θαλάσσια διάσταση της ΚΕΠΑ. Και θεωρώ ότι υποβάλλει κάποιες προτάσεις πολύ αμφισβητούμενες. Thank you very much. And Mrs. please. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Λέζινγκ. Εγώ θα μιλήσω στη δική μου γλώσσα. Και για μας την ΓΚΟΕ υπάρχουν πολλά στοιχεία διαφωνίας, πιο πολλά διαφωνίας παρά σύμπνοιας με τη γενική γραμμή αυτής της ε, έκθεσης. Κάτι το οποίο δεν νομίζω θα σας εκπλήξει. Εν γέννη, νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς ότι αυτή η έκθεση είναι μια συνολική αντιμετώπιση αλλά που έχει σαν στόχο την επέκταση της στρατιωτικής διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έλεγα και οδηγεί και στην στρατικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως είπε και ο κύριος ε, Μπουτικόφερ μια προσπάθεια να δοθεί μια υπέρμετρα ασφαλίτικη διάσταση στην εξωτερική πολιτική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή να ξεπεράσουν όλα τα άλλα θέματα εκτός από την από τη γη της ασφάλειας. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι αναφέρονται όλα τα στρατιωτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τονίζεται ιδιαίτερα η συνεργασία στρατιωτικής, στρατιωτικών πολιτικών αρχών, η ρήτρα ε, αμοιβαία αλληλοβοήθειας κτλ. Ε, και κύριε Γκόμες, ίσως θα πρέπει να μην ξεχάσετε και την πτυχή της ε, ανάπτυξης γιατί αναφέρεστε στα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την λύση των ε, προβλημάτων και αναφέρεστε στη στρατιωτική ε, πτυχή. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει μια καταλήστευση των διεθνών πόρεων επίσης και μια καταστροφή του περιβάλλοντος γιατί αυτά είναι στοιχεία από τα οποία μπορούν να προκύψουν και σειράξεις και εντάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια, η πραγματικότητα είναι ότι όλες αυτές οι συγκρούσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή έχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν συνυπεύθυνο για την έκρηξή τους ή τουλάχιστον σαν κάποιο ο οποίος εκμεταλλεύεται τα αποτελέσματα αυτών των κρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε κάποιο ρόλο στην καταλήστευση του Ινδικού ωκεανού επειδή θέλουμε εμείς να έχουμε ε, αλληλεία ανεξέλεγκτη σε αυτήν την περιοχή που με την επιχείρηση Αταλάντης. Λέτε ότι αντιμετωπίζετε τις πηγές του κακού. Αλλά όλα αυτά τα ξέρουμε ότι προσπαθούμε να χτυπήσουμε τη ρίζα του κακού και στη συνέχεια απλώς ο στόχος είναι να ενισχύσουμε τη στρατιωτική διάσταση και τίποτα άλλο. Αυτή λοιπόν η στρατιωτική διάσταση σχηματοποιείται και γίνεται όλο και πιο συγκεκριμένη σε αυτή την έκθεση. Πρόκειται για προτάσεις, για μια στρατηγική θαλάσσιας ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τις απαραίτητες ενέργειες και τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ανά περιοχές. Θέλω να τονίσω λοιπόν ότι κατά την άποψή μου δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Αυτό είναι θέμα διοκτικών αρχών, αστυνομικών και δικαστικών. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της δημοκρατίας. Ότι κάποιος ο οποίος κάνει ε, εγκλήματα αυτού του είδους θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από κανονικά δικαστήρια και όχι από στρατιωτικές δυνάμεις. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πραγματικά πού βρίσκεται το πρόβλημα. Υπάρχουν προβλήματα όπως η εξασφάλιση των πόρων, η οικονομική εκμετάλλευση που γίνεται προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά για να συγκροτηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένας παγκόσμιος παίκτη στο παιχνίδι εξουσίας. Μια τέτοια επιθετική εξωτερική πολιτική και πολιτική εξωτερικού εμπορίου και η συμμετοχή στον αγώνα για τους παγκόσμιους πόρους και τις πρώτες ύλες, αυτό είναι κάτι το οποίο οξύνει την κλιμάκωση σε στρατιωτικό επίπεδο, σε παγκόσμιο στην παγκόσμιο στίβο. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται τα μεταναστευτικά ρεύματα, αυξάνεται η τρομοκρατία, δεν λύνεται το πρόβλημα της ένδυας και του αποκλεισμού, αλλά οξύνεται ακόμα περισσότερο. Τέλος ένα ερώτημα για τη δημιουργία αυτής της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής που έχετε αναφέρει κυρία Γκόμες. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι αυτή η ακτοφυλακή θα πρέπει να συνεργάζεται με τη Frontex και κατά πόσο όπως εσείς ίσως φαίνεται να προτείνετε, θα πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως με τη Frontex. Έχω λοιπόν τόσες πολλές διαφωνίες και τόσες πολλές αντιρρήσεις με τη γενική κατεύθυνση της εκθέσεως της κυρίας ε, Γκόμες που θα καταλήξω μάλλον να συγγράψω μια έκθεση μειοψηφία για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρος. Κυρία Γκόμες, αν θέλετε να απαντήσετε. Σύντομα παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ για τα σχόλια αυτά, ακόμα και τα πιο επικριτικά σχόλια και προσβλέπω και προς την έκθεση, την εναλλακτική έκθεση που ανέφερε η κυρία Λέζινγκ. Εγώ θέλησα να είμαι φιλόδοξη ακόμα και προκλητική γιατί θέλω να προκαλέσω μια συζήτηση για τα θέματα αυτά. Σίγουρα η έκθεση αυτή βέβαια θα πρέπει να αντανακλά την άποψη της ευρείας ε, πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, ενός ευρέω φάσματος βουλευτών. Και θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο για να εκφράσει την άποψη του Κοινοβουλίου εναντί του Συμβουλίου, το οποίο πρέπει να συζητήσει για το θέμα αυτό. Εγώ φυσικά έχω εκφράσει τις δικές μου απόψεις. Μπορεί να συμφωνεί κανείς, μπορεί να διαφωνεί. Κάποιες πολιτικές ομάδες συμφωνούν, είναι προφανές μαζί μου, αλλά οι απόψεις τους είναι σεβαστές όπως είναι και η δική μου και εγώ θα προσπαθήσω να καταλήξω σε κάποια διατύπωση η οποία οδηγεί σε κάποιους συμβιβασμούς. Τώρα σε, στα σημεία που είναι ιδιαίτερα επίμαχα θα πρέπει να καταλήξουμε στην ψηφοφορία. Αλλά σας υπόσχομαι θα κάνω ό,τι μπορώ για να μπορέσω να συμπεριλάβω όλες τις προτάσεις τροποποίησης και τροπολογιών που θα προέλθουν από τους συναδέλφους. Εγώ πιστεύω ότι είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το εγχείρημα, πολύ χρήσιμο αν θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι. Και θεωρώ ότι ο ρόλος μας θα πρέπει να είναι σαν παγκόσμιου παρόχου ασφαλείας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου, επί τη βάση των ευρωπαϊκών αξιών. Τι νόημα έχει να μιλάμε για την Ευρώπη σαν παγκόσμιο παίκτη <clears throat> όταν δεν έχουμε και μία παγκόσμια ισχύ που περιλαμβάνει και στρατιωτική ισχύ και στον θαλάσσιο τομέα. Νομίζω ότι η προσθέμενη αξία προέρχεται από το να μπορούμε να συνδυάσουμε και τη στρατιωτική και την πολιτική πτυχή και τα αντίστοιχα εργαλεία ώστε να εξυπηρετήσουμε τους στόχους μας που είναι να υποστηρίξουμε τις αξίες μας και τις νομικές αρχές οι οποίες καθοδηγούν πάντα την δράση μας. Επομένως, εγώ... Να σοβαρά όλα όσα μου είπατε, τα σημείωσα, τα έγραψα και αναζητώ ποιες τροπολογίες θα προωθήσω γιατί οπωσδήποτε δεν μπορώ παρά να συμφωνώ με τις προτάσεις ότι θα πρέπει να αναφέρουμε καλύτερα τις εταιρικέ σχέσεις και έχω μια γενικόλογη παράγραφο αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, συγκεκριμένα, να πούμε ποιες εταιρικέ σχέσεις μπορούμε να να προωθήσουμε επίσης. Ο Πολυβρασέλ επέκριναν το ότι έχω ε, λάβει το, το, το, ευρύτερο background της ΚΕΠΑ γιατί ακριβώ γιατί θέλω να δούμε την εμπλοκή μας στα θέματα ασφαλείας παρά τις επικρίσεις πάντως είμαι σίγουροι ότι πρόκειται τελικά να πετύχουμε τη συνένεση. Επίσης, όσον αφορά την ακτοφυλακή και τη Frontex, πρόκειται για ζήτημα επί του οποίου ευχαρίστως να ακούσω τις προτάσεις Γιατί αξίζει να δημιουργήσουν ένα τέτοιο, να συγκροτήσουν τέτοιο σώμα. Να δούμε και πώς θα λειτουργεί, πώς θα συντονίζεται με τη Frontex. Δεν λέω να επεκταθεί παραπέρα από την, τα όσα απασχολούν τη Frontex, αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται από πλευρά οικονομικών πόρων. Αγνοούμε, αγνοούμε τον πλούτο που σημαίνει η θάλασσα. Πολύ σημαντικό αυτό για τα καθημερινά και για τους Ευρωπαίους. Και αυτό επομένω το έχω κατά νου το τον έφερα. Θα ήθελα τώρα. Α, θα ξέρω, ξέρω τι σας προκαλώ. Εκεί που προτείνω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τι γίνεται με κάποιες ε, διευκολύνσεις όπως οι βάσεις των Αζωρών. Πρόκειται για έδαφος ευρωπαϊκό. Είναι, είναι η χώρα την οποία προέρχομαι. Και χρησιμοποιούν τώρα αυτές τις βάσεις οι Αμερικάνοι. Μα γιατί, γιατί, γιατί να μην υπάρχει διμερής εκμετάλλευση. Μιλάμε για πολύ στρατηγικό σημείο γιατί έχουμε τόσο πολλά να αντιμετωπίσουμε στον Ατλαντικό. Το ίδιο ισχύει και για το πράσινο ακροτήριο. Τι γίνεται, τι κάνουν οι άλλοι δηλαδή η Κίνα. Σχεδιάζουν να φτιάξουν αυτικέ βάσει εκεί. Εμεί γιατί μην κάνουμε. Φυσικά επί τη βάση κάποιων ε, συμφωνιών. Μιλάμε για χώρα εκεί, για χώρα εταίρο και είμαι βεβαία ότι θα υπάρχουν και άλλοι και άλλοι και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Α είμαστε επομένω ανοιχτόμυαλοι, γιατί υπάρχουν πολλέ ευκαιρίε. Και δεν θα λέω τώρα για το εμπόριο που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μιλώ για ένα σωρό άλλε προκλήσει που αφορούν την ασφάλεια. Αφορούν την Ένωση, του Ευρωπαίου. Είδατε τι εξάπλωση έχει γνωρίσει η πειρατεία στον Ατλαντικό. Όλα ένα και περισσότερο έχουν εντοπίσει μια τέτοια πραγματικότητα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το εμπόριο. Αφορά και την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Δεν αφορά μόνο τα πληρώματα. Και τους επιβάτες και λοιπά. Γι' αυτό σας λέω να είμαστε φιλόδοξοι. Φιλόδοξοι. Και να μην προδικάζουμε την αντιμετώπιση κάποιων προκλήσεων που γίνονται όλο ένα και πιο ισχυρές. Τέλος. Όσον βρω τον ειρηνικό, συμφωνώ. Είναι πολύ λεπτή εδώ η διατύπωση. προσοχή στο όσα λέμε αυτή την περιοχή. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να παραμιλήσουμε την περιοχή αυτή μια που είναι τόσο μακριά. Θέλουμε ή δεν θέλουμε να είμαστε παγκόσμιου παίκτε, παγκόσμια δύναμη. Τι θα κάνουμε για την ασφάλεια των πολιτών μας και τα συμφέροντά τους και λοιπά θα πρέπει να ζητήσουμε να τα φροντίσουν οι Αμερικανοί. Όχι. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Για να άλλοι προετοιμάζονται για προβλήματα, γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς. Άρα, ας βρούμε την πιο διπλωματική δυνατή διατύπωση, την πιο δόκιμη, την πιο ορθή. Ο κ. Μπουτικόφερ εκτός μικροφώνου. Αν θέλετε να υποτίθεται κάτι τέτοιο, τότε αφήστε αυτή τη διατύπωση, λέει ο κ. Μπουτικόφερ. Ω, πολύ πολύ με ενδιαφέρει επομένω να δούμε τι γίνεται με τις προτάσεις που έχετε. Και όσον αφορά τις περικοπές στην πολιτική άμυνα, συμφωνώ, δεν είμαι κατά των περικοπών κάθε αυτών. Αλλά οι συνέπειές τους είναι το πρόβλημα. Χάνουμε σε δυνατότητες. Και χάνουμε και θέσεις απασχόλησης. Πώς θα το βλέπω οικονομίστηκα το πράγμα. Πρέπει να έχουμε αυτάρκεια στις βάσεις. Μην παραλείπουμε το θέμα. Μην παραμελούμε μάλλον, συγγνώμη, το θέμα. Αυτό που σήμερα. Διότι, συχνά, αυτό το οποίο γίνεται είναι να βλέπουμε αυτές τις δυνατότητες μας, οι ε, πολιτικές, ταχυτικές, σε μερικές χώρες να τις επιμελούνται και σε άλλες να τις παραμελούν. Και γι' αυτό σας λέω. Ας κάτσουμε να το δούμε λογικά. Ας έχουμε μπούσολα ό,τι θεωρούμε αναγκαίες δυνατότητες για το μέλλον μας. Σας ευχαριστώ πολύ, πλέον Πρόεδρος. Και ευχαριστώ και όλα τα σχολεία, Συνεχίζει η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω ότι οι τροπολογίες κατατίθενται μέχρι 22 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Για να είστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Διοργανώνεται και στις 19 Μαρτίου ακρόαση της Επιτροπής μας. Στα 19 Μαρτίου λοιπόν η ακρόαση και μετά μέχρι τις 22, τρεις μέρες ακόμα στη διάθεσή σας για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ και περνάμε στα επόμενα θέματα, πολύ σημαντικά. Εξαγωγή όπλων στο πλαίσιο της κοινή θέση του Συμβουλίου. Όπως ξέρετε, νομίζω ότι είμαστε ο κατά αριθμόν τρίτος ε, μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από κοινού και πολλές ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στην κορυφή του καταλόγου μετά της ε, ΠΑ και τη Ρωσία. Το θέμα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να εναρμονίσουμε τις εξαγωγές των όπλων κάπως, να, υπάρχει, να υπάρχουν καλύτερα πρότυπα, καλύτερες προδιαγραφές. Να δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Λόζινγκ. Θα μιλήσω και πάλι στη δική μου γλώσσα, λέει η κυρία Λούζινγκ. Σας προειδοποιώ για να βάλετε τα ακουστικά σας. Θα ήθελα να σας διορθώσω δεν είμαστε ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, χωρίς το σχετικό κείμενο, θεωρώ ότι δεδομένη της αύξησης των εξαγωγών όπλων και της διάστασης που ενέχεται είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου αποτελεσματικό και ελπίζω να μην υπάρξουν διαφορές σε ό,τι αφορά τις απόψεις που επικρατούν σχετικά με το θέμα αυτό, σε ό,τι αφορά και την κοινή θέση που ψηφίστηκε το 2008, σε ό,τι αφορά την εξαγωγή ε, στρατιωτικού εξοπλισμού και στρατιωτικών τεχνολογικών ε, προϊόντων να υπάρξει ένας αποτελεσματικός έλεγχος από... Στην έκθεση μου λοιπόν προσπάθησα να κάνω συγκεκριμένες προτάσεις για να α, διατυπωθεί στην πράξη αυτή η κοινή θέση και να υπάρξει μια κοινή εφαρμογή. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η κοινή θέση ελήφθησε και εγκρίθηκε βάσει ομοφωνίας. Δεν θέλω λοιπόν από κοινού να να ξανασυζητήσουμε την κοινή θέση, αλλά να τη μεταφράσουμε σε συγκεκριμένα μέτρα. Θεωρώ ότι βασικά θα πρέπει να ενδυναμώσουμε εν γέννη τα θέματα εφαρμογής των κριτηρίων που υφίστανται και θεωρώ ότι να κοιτάξουμε ιδιαίτερα το θέμα του ελέγχου των ε, μέσων πολιτικού, των πολιτικών προϊόντων, μέσων πολιτικής ε, άσκησης της φύσης. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βελτιωθούν ε, οι εθνικές ε, μέθοδοι συλλογής στατιστικών στοιχείων και εναρμονισμός. Η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου έχει συμβάλει ασφαλώς σε θέματα τυποποίησης, αλλά αυτά δεν επαρκούν. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν πλήρη στοιχεία τυποποιημένα από όλα τα κράτη-μέλη προκειμένου να υπάρχει χρήσιμη και ρεαλιστική αξιολόγησή τους. Θα πρέπει να έχουμε και πιο πολλές πληροφορίες στη διάθεσή μας, ε, όπως για παράδειγμα απαρίθμηση των χωρών προς τις οποίες δεν πρέπει να γίνονται και δεν επιτρέπεται να γίνονται εξαγωγές βάσει ποιου κριτηρίου και Επίσης, πιο πολλές πληροφορίες σε σχέση με το πού καταλήγουν ε, τα όπλα. Επίσης, συμπερίληψη της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών κοινοβουλίων ως ανεξάρτητοι παράγωγοι, παράγοντες ε, ελέγχου. Και τέλος, θα ήθελα να τονίσουμε και την διεθνή διάσταση του προβλήματος αυτού και γι' αυτό αναφέρω και την ε, συνθήκη για το εμπόριο όπλων. Ανέφερα τα σχετικά ζητήματα στην έκθεση δεδομένης και της διάσκεψης του ΟΗΕ τον Μάρτιο σε θέματα εξαγωγής όπλων. Θα ήθελα να προσθέσω ότι θα καλωσόριζα ένα τέτοιο σύστημα ελέγχου δεσμευτικό ακόμα και αν σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να τύχει διαπραγμάτευσης από τις χώρες. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο ζήτημα που αναφέρω στην έκθεσή μου για την ε, μετατροπή και τη μείωση του εξοπλισμού. Γνωρίζω ότι το θέμα τα μετατροπής ε, κυρίως είναι θέμα κοινωνικό πάνω απ' όλα και πολύ φοβάμαι ότι ρεαλιστικά το κοινοβούλιο αυτό δεν θα υποστηρίξει την ε, τοποθετησή μου, αλλά είμαι απόλυτα απεπισμένη ότι αυτό αποτελεί κάτι το απολύτως απαραίτητο και θεωρώ στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί κάτι που είπε ο κύριος Μπουτικόφερε ή έχουν γίνει έρευνες για το ποιος είναι ο ρόλος ε, των ε, όπλων και διαπιστώνεται ότι ένα δολάριο για την παραγωγή όπλων και ένα δολάριο για τον τομέα Τη κοινωνική ανάπτυξη αποφέρει το δολάριο στην κοινωνική ανάπτυξη τρεις φορές πιο πολλέ θέσει εργασία. Κλείνω λοιπόν λέγοντα αυτό το αναφέροντας αυτό το στοιχείο. Ευχαριστώ κυρία Λούζιν και θα πάρω εγώ το λόγο γιατί είμαι σκιώδη είσαι από το ΕΛΚ. Θα μιλήσω πολωνικά. Ευχαριστώ. Είναι ένα πρόβλημα λοιπόν το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και σημαντικό το οποίο ε, αναφέρεται στην έκθεσή σας κυρία Λέζινγκ. Εγώ συμφωνώ με την ε, δομή της έκθεσης. Έχω να κάνω βέβαια ορισμένε παρατηρήσεις. Κάποιες μπορεί να είναι πιο σημαντικές από τις υπόλοιπες, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση οι ισχυώδεις μαζί σας κυρία Λέζονγκ. Είμαι πεπισμένος ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι θετικό για όλους. Συμφωνώ για το γεγονός ότι η έκθεση αυτή διαλαμβάνει και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική η οποία δεκρίθηκε το Δεκέμβριο και, και εσείς κυρία Λέζινγκ το υπογραμμίσατε ότι υπήρξαν πέντε κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τρομοκρατία, όπλα μαζικής καταστροφής, περιφερειακές σειράξεις, κατάρρευση ορισμένων κρατών και οργανωμένη εγκληματικότητα. Επίσης υπάρχει το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας συμβατικών όπλων που συνδέεται με αυτές τις πέντε προκλήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει έλεγχος των εξαγωγών όπλων. Το κύριο κείμενο το οποίο αναφέρεται είναι η κοινή θέση του Συμβουλίου η οποία διαμορφώθηκε το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους και αφορά τον στρατιωτικό εξοπλισμό και τα όπλα εν γέννη. Στρατιωτικού χαρακτήρα. Είναι μια θέση η οποία είναι επικαιροποιημένη και είναι ένα εργαλείο το οποίο ξεπερνάει όλα αυτά τα εργαλεία που είχαμε στο παρελθόν. Μας επιτρέπει να έχουμε ένας σε βάθος έλεγχο των ε, εξαγωγών οπλικών συστημάτων όταν υπάρχουν διαμετακομίσεις, χρήση ενδιαμέσων, μεταλαμπάδευση τεχνολογίας. Θέλουμε λοιπόν να εναρμονίσουμε πλήρως την πολιτική εξαγωγών των κρατών μελών. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος τώρα, σε ορισμένα σχόλια τα οποία αφορούν το σχέδιο εκθεσή σα. Φυσικά, θα σας δώσω και όλα αυτά τα στοιχεία εγγράφως. Θα καταθέσω και τροπολογίες στην εκθεσή σας. Πρώτα απ' όλα όμως για τις αιτιολογικές σχέσεις σκέψεις έχω κάποια σχόλια τα οποία θέλω να διατυπώσω για τις παραγράφους του κειμένου. Γιατί αναφέρεστε ήδη σε στοιχεία τα οποία λειτουργούν στην πραγματικότητα με την ε, ενίσχυσή τους μπορούμε να έχουμε μάλλον με την ε, χρήση αυτών των στοιχείων μπορούμε να μειώσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής εξοπλιστικής βιομηχανίας. Πιστεύω επίσης ότι στην πρότασή σας αναφέρετε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει κάποιος μηχανισμός για τον συντονισμό των πολιτικών εξαγωγής, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες μέθοδοι ανταλλαγής πληροφοριών, υπάρχουν συστήματα κοινοποιήσεων. Όταν δίδονται εξαγωγικέ άδειε, υπάρχει κοινοποίηση στα άλλα κράτη-μέλη. Επομένω, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο έλεγχο των εξαγωγών όπλων, επίση. Έχει σαν στόχο να μην ενισχύσει την τρομοκρατία. Είναι λοιπόν τέτοιε ρήτρε οι οποίε ε, διέπουν τι εξαγωγέ αυτέ που ισχύουν ήδη σήμερα. Και έρχομαι στην τελευταία παράγραφο τη έκθεσή σα. Εδώ πρέπει να είμαστε λίγο πιο μετρημένοι. Ιδίω για τα θέματα ανταγωνιστικότητα που ανέφερα προηγουμένω, αλλά λαμβάνοντα υπόψη και την τωρινή κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις περιφερειακές σειράξει που σοβούν, με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και της Βόρειας Κορέας, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με όλε τι ανησυχίε που έχουμε για συγκεκριμένε περιφερειέ και περιοχέ του κόσμου. Αυτά δεν πρέπει να επηρεάσουν υπερβολικά και υπέρμετρα τις ε, εξοπλιστικές βιομηχανίες των χωρών μας. Αλλά έχουμε και υποχρέωση οι οποίες απορρέουν από τη συμμετοχή των χωρών μας στο ΝΑΤΟ. Και αυτό πρωτού σκεφτούμε καν τι κάνουν χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της εταιρικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και τη συνεργασία του ΝΑΤΟ με τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να θυμηθούμε τι είπε το Μάιο του 2012 ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει ένα παγκόσμιο παίκτη, θα πρέπει ήδη από σήμερα να βρει τι δυνατότητε εξυγχρονισμού και ανάπτυξης ορισμένων βιομηχανικών κλάδων που άπτονται των εξοπλισμών. Για να γίνουν λοιπόν όλα αυτά υπάρχει μια πτυχή απαράγραπτη που είναι ο έλεγχος των εξοπλισμών. Σας ευχαριστώ. Και δίνω το λόγο στην κυρία Κοπά τώρα. Like Mrs. Να συγχαρώ την κυρία Λόζινγκ για την ε, εκθεσή της. Καλύπτει όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της κοινής τη 2008 για την εξαγωγή των όπλων. Θα θέλουμε να πιστεύουμε ότι γενικά το θέμα αυτό δεν θα μας ε, διαιρέσει διότι επί πολλά έτη θέλουμε να ε, προσαρμοστεί αυτή η κοινή θέση και ότι θα πρέπει τελικά να υπάρχει ένα δεσμευτικό νομοσχέδιο, κάποιου ε, κοινά πρότυπα, κοινού κανόνε που να καλύπτει την στρατιωτική τεχνολογία και εξοπλισμό. Ο, ο έλεγχο των, εξ, των εξαγών θα πρέπει να συμπληρώσει άλλε διαστάσει τη εξωτερική μα δράση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πρόληψη και διαχείριση των κρίσεων, αλλά και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκόσμια και ακριβώς όπως λέει και η συγγήτρια. Όταν έχει τη ώρα τη εφαρμογή όμω, επιδέχονται μεγάλη βελτίωση στα πράγματα. Τα 8 κριτήρια τη κίνηση θέση δεν έχουν ληφθεί σοβαρά από πολλά κρατημέλη και επομένω τα οικονομικά συμφέροντα κυριαρχούν. Και γι' αυτό το μήνυμα θα πρέπει να είναι δυναμικό να τονίζουμε την ιδιαίτερη ευθύνη των χωρών που παράγουν όπλα σχετικά με αυτά που είπαμε. Η έκθεση επίσης τονίζει που είναι τα κενά όσον αφορά ε, τον έλεγχο τη εφαρμογή και τα κριτήρια τη εφαρμογή. Προτείνει να υπάρχει μια πρώτη τυποποιημένη ε, μέθοδος ελέγχου, να εμπλέκεται και το Κοινοβούλιο, γύρω των Πολιτών και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα του κανόνε που διέπουν τα αγαθά διπλής χρήσης και πρόκειται για κάποιες κυρώσεις για περιπτώσεις παραβάσεων, οπότε κατά την άποψή μου και της πολιτικής μου ομάδας είναι σημεία από τον οποίο συμφωνούμε όλα αυτά, όμως δεν θα πρέπει να είμαστε παντού αρνητικοί γιατί θα πρέπει να εγκρίνουμε μια κοινή θέση η συγκρότηση της ομάδας εργασίας και επίσης αναθεωρημένη ε, μορφή του κειμένου, αυτό που το λέμε οδηγίες χρήσης, όλα αυτά ορθά λέγονται στην ε, έκθεση επίσης στην ε, έκθεση της ΚΟΑΜ του Δεκεμβρίου αναγνώσει το Συμβούλιο ότι θα πρέπει να ε, επεξεργαστούμε περαιτέρω την κοινή θέση η δε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ως σκοπό να υποστηρίζει τις προπαθίες αυτές και να προχωρήσουμε προς πλήρη εναρμόνιση των πολιτικών των εθνικών για τις εξαγωγές και επί τη βάση των δικών μας και παγκοσμίων αρχών οπότε οι έλεγχοι μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικοί εάν ισχύσουν και εφαρμοστούν με τρόπο συνεπή, ομοιόμορφο παντού παγκοσμίω. Οπότε ευχαριστούμε την εισηγήτρια, την κυρία Λόζιν, γιατί έχει ένα κεφάλαιο εδώ για τις διεθνείς ε, αποφάσεις που οδηγούν σε μια τέτοια υγιή πολιτική για την εξοχή των όπλων. Τέλος. Εμείς ελπίζαμε άλλως να έχουν τα πράγματα. Δεν ε, οδηγηθήκαμε σε κάποια λύση πριν τις διαπραγματεύσεις της Νέας Υόρκης τον επόμενο μήνα. Άρα, θα πρέπει να επαναλάβουμε την ολοκληρωτική μας υποστήριξη των προσπαθειών. Εάν δεν πάνε καλά διαπραγματεύσει, θα πρέπει στην έκθεση να καλύψουμε την κατάληξη αυτών των διαπραγματεύσεων. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γετμακή. Ευχαριστώ. Και θα συνεχίσω στα φιλανδικά. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Λεωζίν για μια πολύ συνεκτική έκθεση, ένα σχέδιο έκθεσης και εκ τον τονίσω ότι σήμερα παρά το γεγονός ότι διάβασα γρήγορα, γρήγορα την έκθεση, δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες και λεπτομερείς σχόλια. Είμαι βέβαιη ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό αργότερα. Και θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες για να συνεργαστούμε. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποια από τα στοιχεία που περιλαμβάνει η έκθεση. Νομίζω ότι Σωστά τονίζετε ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου σε ό,τι αφορά την εξαγωγή των όπλων. Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν βάσει της κοινή θέση. Αυτό δεν γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις σήμερα. Επίσης, στην έκθεση περιλαμβάνεται το ερώτημα του πώς μπορούμε να αλλάξουμε την αντιμετώπιση μας. Γιατί δεν αρκεί. να αλλάξουν κάποια επιμέρους ζητήματα. Πρέπει να αλλάξει η όλη νοοτροπία μας. Αυτό ίσως είναι και ελαφρώς διαφορετικό ζήτημα. Προς την εισηγήτρια. Να τονίσω της, ε, στη σημασία της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Άμυνας δημιουργεί θέσεις εργασίας και είναι θεωρώ σημαντικό η Ευρώπη να έχει έναν τέτοιο κλάδο. Αυτό θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε περαιτέρω και την τεχνολογία μας ασφαλώς. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια τεχνολογία παντού εκτός από την Ευρώπη. Ιδάλλως θα φύγουν αυτές οι δουλειές από την Ευρώπη. Και είναι η αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι έχουμε και αγορά για τα όπλα αυτά κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Μέση Ανατολή, στην Βόρεια Αφριοκή. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποιους κανόνες για το πώς θα πολλούνται όπλα σε αυτές, ε, σε αυτές τις χώρες. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν αλλαγή νοτροπίας, θα πρέπει να υπάρξει και ανάληψη των ευθυνών μας σε ό,τι αφορά τον ορισμό των κανόνων αυτών. Ασφαλώς, αυτοί που φέρουν την ευθύνη είναι αυτοί που δίνουν την τελική ε, άδεια για την εξαγωγή των όπλων. Οι κυβερνήσει μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ελέγχει την εφαρμογή των σχετικών κανόνων. Θα πρέπει να δραστηριοποιούμαστε πάντα γρήγορα όταν ε, ο έλεγχος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν εφαρμόζονται οι αρχές μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Κρονμέρκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως είπαν και οι άλλες ε, ομάδες, καλωσορίζουμε και εμείς την εκθεσή αυτή. Έχουμε κάποια μικρά σχόλια τα οποία θα τα διαβιβάσω στην κυρία Λούζινγκ. Τρεις τομείς ωστόσο υπάρχουν στους οποίους θα θέλαμε προτάσεις της εισηγητρίας. Καταρχάς, η πρόταση για να υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος. Θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρχουν και κάποιες εναλλακτικές ιδέες για το πώς θα βελτιωθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Κατά δεύτερον, στην παράγραφο 7 υπάρχει ένα πολύ ουσιώδες σημείο που αναφέρει ότι δεν υπάρχει έλεγχος κατά πόσον πληρούνται τα οκτώ κριτήρια και ότι δεν υπάρχει μηχανισμός επιβολής κυρώσεων. Πολύ βασικό αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να διαπιστώνουμε κατά πόσο πληρούνται και ακολουθούνται τα κριτήρια που έχουν τεθεί και να υπάρχει και δυνατότητα επιβολής κυρώσεων. Και πάλι λοιπόν θέλουμε προτάσεις από την εισηγήτρια για το πώς θα μπορέσουμε να κινηθούμε στην κατεύθυνση αυτή στην τρέχουσα έκθεση προόδου, ετήσια έκθεση προόδου, αναφέρεται ότι κάποιες χώρες δεν αναφέρουν τι έχουν εξαγάγει χώρες όπως το Βέλγιο, η Ελλάδα και άλλες. Νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και θα πρέπει να κατατεθούν και πάλι συγκεκριμένες προτάσεις. Τέλος, εντοπίζω δύο τομείς στους οποίους θα θέλαμε να υπάρχει γενική πρόοδος. Καταρχάς, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σημαντική πτυχή για το Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε πιο συγκεκριμένη σύνδεση μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εξαγωγής όπλων. Κατά δεύτερον, πριν τα πρινικά ζητήματα του Ιράν και της Βόρειας Κορέας, αναφέρεται και στην έκθεση, υπάρχει αύξηση των πωλήσεων περινικού εξοπλισμού ευαίσθητου. Θα πρέπει κάπου να τονίσουμε ότι δεν είναι δυνατό να συνεχίσει αυτό και δεν είναι αποδεκτό και ότι τα, η τεχνολογία, η πυρηνική τεχνολογία η ευαίσθητη θα πρέπει να περιορίζεται. Ευχαριστώ. Κύριο Τέρχο, τελευταίος εισηγητής μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Εγώ είδα μόλις αυτή την έκθεση, δεν είχα το χρόνο να τη διαβάσω προσεκτικά. Η κοινή θέση του Συμβουλίου παρουσιάζει στοιχεία τα οποία εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν και να εφαρμοστούν ομοιόμορφα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια κοινή κατεύθυνση και να έχουμε συμφωνία μεταξύ μας για το πώς θα μπορέσουν όλα αυτά τα κριτήρια να γίνουν κατανοητά με ενιαίο τρόπο και να εφαρμοστούν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαι τόσο σίγουρος για ορισμένα άλλα θέματα μέσα στην έκθεση αυτή. υπάρχει το θέμα του ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για, όλα αυτά, για όλες αυτές τις ενέργειες. Η εισηγήτρια δίνει την εντύπωση ότι θεωρεί αρνητικό το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει όλα αυτά τα οπλικά συστήματα. Νομίζω πρέπει να το δούμε από τη θετική του πλευρά. Υπάρχει και η επικεφαλίδα αφοπλισμός στην έκθεση αυτή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της έκθεσης. Αναφέρεται στην παράγραφο 27, στην τελευταία φράση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μετατρέψει την εξοπλιστική βιομηχανία από την παραγωγή εξοπλιστικών συστημάτων σε πολιτικού χαρακτήρα παραγωγή, αλλά δεν ξέρω πώς θα μπορέσετε να το κάνετε αυτό στην πράξη. Είναι δύσκολα λοιπόν όλα αυτά να τα πει κανείς σε δύο λόγια. Νομίζω πρέπει να συζητήσουμε λίγο περισσότερο για το θέμα αυτό. Καταλαβαίνω όμως ότι υπάρχουν και κάποια πολύ χρήσιμα θέματα στην έκθεση και περιμένω τη συζήτηση με την ε, εισηγήτρια. Υπάρχουν τρεις ακόμα που πρέπει να λάβουν το λόγο. Δίνω το λόγο στην κυρία Γκόμιση πρώτα. Δεν έχω σοβαρές διαφωνίες με την κυρία Λόζιν. Είναι μια χρήσιμη έκθεση. Θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω αν είναι πιο λεπτομεριακά τα παραδείγματα που δίνει η κυρία Λέζιν. Όσο πιο πολύ υπογραμμίζουμε τις αντιφάσεις ανάμεσα στις δηλώσεις και τις πράξεις των κρατών μελών μας και τον μη σεβασμό λοιπόν των ε, κριτηρίων που διατυπώνουν. Αυτό νομίζω ότι είναι χρήσιμο που κάνει η συγγήτρια και όπως είπε και για την κυρία Κρόνμπεργκ. Πιστεύω ότι όταν μιλάμε για τεχνολογίες επισκόπησης και παρακολούθησης αυτά και όταν λέτε ότι αυτά δεν περιλαμβάνονται στον κοινό κατάλογο οπλικών συστημάτων, θα ήταν χρήσιμο να έχετε κάποια παραδείγματα εδώ. Οι χώρες οι οποίες εξήγαν αγαθά στην ε, Λιβύη και άλλες χώρες το οποίο που παραβιάζουν τους κανόνες μας, αυτό πρέπει να τονιστεί. Και εδώ πέρα αναφέρεται και η Τη Λιβύη και τι χώρε Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, παραδείγματο χάρη, που παραβιάζαν του κανόνε. Όλα αυτά πρέπει να υπογραμμιστούν. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή μπορεί να μα δώσει τι λεπτομέρειε που είναι καθοριστικέ και μπορεί να κάνουν τα κράτη-μέλη να τροποποιήσουν τη δράση του. Αν παραμείνουμε σε επίπεδο ιδέων χωρί να δώσουμε λεπτομεριακά στοιχεία, τότε συνεχίζουν τα πράγματα όπω ήταν και στο παρελθόν. Και συμφωνώ σε ότι όλα αυτά τα πράγματα που έχουν να κάνουν με ευαίσθητη ποινική τεχνολογία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση και νομίζω θα ήταν και ενδιαφέρον να δούμε και ποιο είναι και ο αντίκτυπο τη κρίση στον τρόπο με τον οποίο τα δικά μα κράτη-μέλη αντιμετώπισαν όλα αυτά τα τόσο ευαίσθητα θέματα παραγωγής πολεμικού στρατιωτικού υλικού και το γεγονός ότι υπάρχουν εξαγωγές τεχνολογιών διτής χρήσης ή και καθαρά στρατιωτικού χαρακτήρα σε χώρες που θα έπρεπε να αποκλείονται βάσει των κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί από το Συμβούλιο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκθεση λοιπόν για να τονίσουμε αυτό το στοιχείο. Ευχαριστώ πολύ και ο πρόεδρο, ο κ. Κάμπελ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εν συντομία, πολύ φοβάμαι ότι είμαι αντίθετο σε αυτή την έκθεση. Μου φαίνεται ότι πρόκειται για α, αναφορά σε κάποιες πολύ σημαντικές ε, βιομηχανίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία των όπλων στην Ηνωμένο Βασίλειο και στη Σουηδία και αλλού. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κοινή θέση. Χρειάζεται να είμαστε όλοι μας υπεύθυνοι. Για παράδειγμα στο 12, γιατί τα κρατημέλη θα πρέπει να παρέχουν ε, ε, λεπτομερείς αναλύσεις των εξαγωγών τους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι ε, αποδεκτό και αποτελεί παραβίαση της επικυριαρχίας. Είμαι κατά της έκθεσης. Συγγνώμη, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Αφοκλέους. Καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την προσπάθεια που κατέβαλε που πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη και βέβαια το σχόλιο της η καλύτερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλος στον κόσμο είναι μια διόρθωση με πολλαπλά μηνύματα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πολλές θέσεις εργασίας βρίσκονται στον ευρωπαϊκό χώρο. Πολλά κέρδη και πολιτισμός αναμένεται να υπάρχει. Συμφέροντα βιομηχανιών αλλά και βεβαίως κρατών στον ευρωπαϊκό χώρο. Νομίζω ότι σαν θέση αρχής όλοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να μειώνονται οι εξοπλισμοί στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια. Να έχουμε πληροφορίες που καταλήγουν από την Ευρώπη αλλά και από τις Ηνωμένε Πολιτείε και τη Ρωσία και άλλες χώρες. Να υπάρχει ένας έλεγχος για όλους και νομίζω αυτό πρέπει να είναι και το πολιτικό μήνυμα που πρέπει να εκφράσουμε. Η δική μου ερώτηση είναι η εξής. Με ποιον τρόπο, με ποια μεθοδολογία θα μπορεί να γίνεται πρακτικά αυτός ο έλεγχος. Ακόμα ο εξοπλισμός των περιορισμών και βεβαίως μέσα από την εισήγηση η οποία πρέπει να προσθέσει εκτιμώ εγώ θα πρέπει να λαμβάνεται πάρα πολύ σοβαρά υπόψη αυτό που ήδη έχω αναφέρει ότι όποια προσπάθεια καταβάλλεται γίνεται, διορθώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει στο μυαλό μας να βρίσκεται η ανταγωνιστική σχέση είτε μας αρέσει είτε όχι με άλλες χώρες περιορίζουμε να αναφέρω δύο οι Ηνωμένε Πολιτείε και Ρωσία σε αυτόν τον τομέα. Γι' αυτό χρειάζεται νομίζω, πιστεύω και κλείνω μια πρόσθεση στην εισήγηση με περισσότερη λεπτομέρεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κρόμπερκ ήθελε να προσθέσει κάτι. Διαδικαστικό σχόλιο. Πήραμε την έκθεση μόλις σήμερα και η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 6 Μαρτίου. Λίγο περισσότερο χρόνο μάλλον θα χρειαζόμαστε για τις τροπολογίες. Εντάξει, θα το ελέγξουμε με τη γραμματεία. Και εγώ να κάνω ένα σχόλιο για την, ε, τις εκθέσεις για τις εξαγωγές όπλων. Πολλές φορές έχουμε μια κατάσταση που παράγονται τα οπλικά συστήματα σε μια χώρα, αλλά πολλούνται από μια εταιρεία που βρίσκεται σε μια άλλη χώρα. Έχουμε παραγωγικά την Αμερικανική εταιρεία Sikorsky, η οποία παράγει ελικόπτερα στην Πολωνία και εξάγονται στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά το θέμα είναι αν είναι αμερικανικές εξαγωγές ή πολωνικές εξαγωγές μέσω αυτού του εργοστασίου. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα σαφή. Κυρία λέζου θέλετε να κλείσετε τη συζήτηση. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Όλα αυτά τα σχόλια λοιπόν είναι σχόλια τα οποία εγώ πρέπει να κατατάξω σε σχόλια τα οποία είναι γενικά κατά της κατεύθυνσης της έκθεσης ή που εν πάση περιπτώσει εκφράσουν πάρα πολλές ανησυχίες και αμφισβητήσεις και αυτά τα σχόλια τα οποία έχουν σαν στόχο μια βελτίωση της έκθεσης και, μια, και ένα εμπλουτισμό της. Εγώ θα ήθελα να σκεφτώ να αντιμετωπίσω καταρχήν αυτά που εκφράσουν αρνητικές σκέψεις ή αντιρρήσεις. από τη δική μου οπτική γωνία, εγώ πιστεύω ότι έχουμε την κοινή θέση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν, λοιπόν, η έκθεσή μου αμφισβητεί αυτήν την κοινή θέση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ότι η έκθεσή μου αποτελεί μια διαμφισβήτηση της κοινή θέσης του Συμβουλίου. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτή τη θέση ε, απορρέει το περιεχόμενο της εκθεσής μου. Εγώ θέλω να έχουμε μια διαφορετική συζήτηση για τα θέματα αυτά. Και τονίζω ότι αν δεν μπορέσουμε στο τέλος να καταλήξουμε σε μια αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου επί τη βάση της κοινής θέσης αυτής, τότε όλα αυτά τα οποία προτείνονται από την κοινή θέση θα πρέπει να καταργηθούν. Οι πολίτε Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καταλάβουν περί τίνο πρόκειται για όλα αυτά τα ζητήματα. Κύριε Λίζεκ, έχω παρουσιάσει αυτή την έκθεση ήδη και στο Βερολίνο, όπου υπήρχαν πολύ ενδιαφερόμενοι από τον ε, βιομηχανικό αυτό κλάδο και είναι σαφές ότι υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων για τα θέματα αυτά. Αυτό το οποίο θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η έκθεση της, η πρόθεση αυτής της έκθεσης δεν είναι να περιοριστεί μονάχα στο εμπόριο όπλων. Ο στόχος αυτής της έκθεσης είναι να αντιμετωπιστεί το εμπόριο όπλων το οποίο παραβιάζει τα κριτήρια της ε, του Συμβουλίου και να δούμε το πώς μπορούμε να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο. Και για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουν τα πράγματα και αυτό είναι μια συζήτηση που αρμόζει σε μια κοινωνία και είναι συζήτηση επί των αξιών μιας κοινωνίας που θα πρέπει να καθορίσει κατά ποιε συνθήκες μπορεί να λειτουργεί η, η εξοπλιστική βιομηχανία και αν μπορεί να προσπορίζεται υπέρμετρα κέρδη από εξαγωγές σε χώρες όπου καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι λοιπόν μια πολιτική συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει και η οποία δεν περιοριστεί μονάχα στην εκθεσή μου. Αυτά τα οποία είπε η κυρία Γκόμες. Κυρία Γκόμες, αυτό το οποίο ζητάτε δεν στρέφεται κατά της έκθεσης, γιατί η έκθεση αυτή δεν αφορά την πρακτική του εμπορίου όπλων. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει για μένα αυτό θα μπορούσε να είναι ένα παράτημα. Μια τέτοια εξ, ε, εξέταση. Εγώ ξεκινώ από το γεγονός ότι πολλούνται όπλα σε χώρες όπου παραβιάζονται τα κριτήρια για την εξαγωγή όπλων, παραγωγικά στη Σαουδική Αραβία, στη Λιβύη. Και από αυτές τις ενέργειες εγώ καταλήγω στο συμπέρασμα ότι τα κριτήρια και η εφαρμογή αυτών των κριτηρίων δεν γίνεται με ένα αποτελεσματικό τρόπο. Δεν θέλω λοιπόν να αλλάξουμε τελείως το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης. Κυρία Κρόνπερκ, εσείς λέτε ότι ότι θα ήταν χρήσιμο να έχουμε περισσότερες πληροφορίες, ε, πιο λεπτομεριακές πληροφορίες. Ίσως δεν κατάλαβα τώρα ακριβώς τι εννοούσατε. Μπορούμε να το συζητήσουμε μετά διμερός. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι λέμε όταν μιλάμε για χώρες στις οποίες χρησιμοποιούνται τα εξαγόμενα όπλα για να κατασταλούν οι ελευθερίες και να καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τη βάση αυτή τη συζήτηση μπορούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με ποια μορφή μπορεί να υποβάλει προτάσεις προς τα μεμονωμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Γιαχτεμάχη, είπατε ότι πρέπει να υπάρξει μια μεταστροφή στην κολτούρα του εμπορίου όπλων να έχουμε μια μεγαλύτερη υπευθυνότητα, ναι, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι επαρκές. Αυτό φαίνεται και από τις περιπτώσεις χωρών όπως η Σαουδική Αραβία και η Λιβύη που στη συνέχεια τα όπλα τα οποία παίρνουν μπορούν να τα μεταφέρουν σε τρίτες χώρες ή να τα πουλούν σε τρίτες χώρες. Είναι απαραίτητο να έχουμε διαφάνεια, αλλά για αυτούς οι οποίοι παραβιάζουν τους κανόνες δεν αρκεί η διαφάνεια θα πρέπει να έχουμε και τρόπους με τους οποίους θα επιβάλλουμε κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων. Οι επιπτώσεις για την εξοπλιστική βιομηχανία δεν τα ανέφερα αυτά ήδη. Θα πρέπει να σκεφτούμε και πάλι ότι πάρα πολλά πράγματα γίνονται ουσιαστικά εγκρυπτό, γίνονται στο σκοτάδι και εκφεύγουν από κάθε μορφή ελέγχου. Και θα πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Και αυτό φυσικά είναι ένα θέμα που αφορά πολιτικές αποφάσεις. Δεν θα πω τώρα σε όλες τις λεπτομέρειες, θα συζητήσουμε και με τους σχεδόν Πιστεύω ότι πολλά πράγματα μπορούν να τροποποιηθούν στην έκθεση αλλά θέλω να σας πω και πάλι ότι εγώ εστιάζω στα θέματα της εφαρμογής των κριτηρίων και η δική μας δυνατότητα να επηρεάσουμε τα πράγματα είναι αρκετά περιορισμένη. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ερχόμαστε στο επόμενο θέμα, η κατάσταση των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δομών και οι μελλοντικέ ε, ε, προοπτικές. Έχει το λόγο η κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξωτερικές της δράσεις σε σχέση με άλλους οργανισμούς έγκυται στη μοναδική της δυνατότητα να μπορεί να κινητοποιεί ένα πλήρες φάσμα πολιτικών, οικονομικών, αναπτυξιακών και ανθρωπίνων μέσων που μπορούν να συνδράμουν στις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων αυτή η συνολική προσέγγιση προσφέρει μια μοναδική ευελιξία και αποτελεσματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι οι στρατιωτικές δομές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της προσέγγισης εφόσον όλα τα άλλα μέσα που έχει στην κατοχή της η Ένωση δεν μπορούν να προσφέρουν τα απαραίτητα αποτελέσματα. Η έκθεσή μου σχετικά με τις στρατιωτικές δομές δηλαδή την τωρινή κατάσταση, τις μελλοντικές προοπτικές, σκοπεύει να εστιάσει ακριβώς σε αυτό το σημείο της συνολικής προσέγγισης. Σήμερα είναι η πρώτη συζήτηση που έχουμε και θέλω να ακούσω και τις ιδέες των συναδέλφων επί του θέματος, πιστεύοντας ότι ο διάλογος θα είναι επικοδομητικός και θα βοηθήσει στην κατάρτιση του τελικού σχεδίου. Θα σας αναφέρω ενδεικτικά το χρονοδιάγραμμα της έκθεσης στις 26 Φεβρουαρίου σήμερα γίνεται η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Στις 12 Μαρτίου θα είναι η τελευταία προθεσμία για να σταλεί προς μετάφραση το κείμενο της έκθεσης. Η 19η Μαρτίου θα είναι η μέρα κατά την οποία θα γίνει πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Η προθεσμία για τις τροπολογίες θα είναι 11η Απριλίου στις 12 η ώρα ε, η δεύτερη συζήτηση επί της εκθέσεως θα γίνει στις 16 Μαΐου. Θα την εγκρίνουμε στην ΑΦΕΤ στις 29 ή 30 Μαΐου και τον Ιούλιο θα έρθει στην Ολομέλεια. Πρέπει να γίνει σαφές από την αρχή ότι η έκθεση δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τη συνολική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε προσπαθεί να υπερτονίσει κάποιες επιμέρους διαστάσεις έναντι κάποιων άλλων. Θεωρώ ότι αυτή η επισήμανση πρέπει να γίνει κατανοητή για να μην εμπλακούμε σε ατέρμονες συζητήσεις για τη φύση της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Βεβαίως στο κείμενο θα γίνουν αναπόφευκτα κάποιες αναφορές και στα μη στρατιωτικά μέσα που έχει στην κατοχή της η Ένωση. Αλλά αυτές θα έχουν καθαρά συμπληρωματικό χαρακτήρα και η χρήση τους θα διευκρινίζει περισσότερο συγκεκριμένες παραμέτρους που έχουν άμεση σχέση με το στρατιωτικό σκέλος. Παρά την εδώ και χρόνια εκπεφρασμένη δέσμευση της Ένωσης για την άσκηση ισχυρής αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής για την ασφάλεια και την άμυνα, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Ένωση στο κομμάτι της ανάπτυξης καθαρά στρατιωτικών ικανοτήτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο επίπεδο των φιλοδοξιών που η ίδια έχει θέσει. Η φιλοδοξία της Ένωσης για σταδιακή διαμόρφωση μιας κοινή αμυντικής πολιτικής εκφράζεται σε επίπεδο συνθήκων και αποφάσεις μας θα έχουν ως γνώμονα την σταδιακή επίτευξη αυτού του στρατηγικού στόχου. Η αυτονομία βέβαια αυτή θα σέβεται τις υφιστάμενες συμμαχίες, ιδίως όσο αφορά το ΝΑΤΟ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε στις προσπάθειες προώθησης μιας στρατηγικής αυτονομίας σε επιχειρησιακό επίπεδο. Σαφέστατα η προσπάθεια αυτή λόγω της οικονομικής κρίσης και των συνεχών περικοπών στους αμυντικούς προϋπολογισμούς γίνεται δύσκολη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό του αμυντικού σχεδιασμού. Οι συνέργειες που μπορούν να επιτευχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να δώσουν τη λύση στα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σημερινό οικονομικό αδιέξοδο. Όσο και αν φαντάζει παράδοξο, η κρίση μπορεί να γίνει ευκαιρία για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, ώστε να γίνουν όλα όσα δεν προχώρησαν σε προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να επανεξετάσουμε τα εργαλεία και τους μηχανισμούς που χρειάζεται η Ένωση για την επίτευξη των δεσμεύσεών της. Η έκθεση που βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο θα κινηθεί στους ακόλουθους άξονες. Πρώτον, στις δομές σχεδιασμού και εκτέλεσης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Δεύτερον, στις δυνάμεις ταχείας αντίδρασης. Τρίτον, στις μόνιμες πολυεθνικές δομές των κρατών μελών. Και τέταρτον, στην ανάπτυξη δομών και ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των σημερινών αδυναμιών. Είναι γεγονός ότι η έλλειψη ενός επιχειρησιακού στρατηγίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων δυσκολεύει πάρα πολύ την ετοιμότητα της Ένωσης. Την εμποδίζει να αντιδράσει αποτελεσματικά και έγκαιρα στην αντιμετώπιση των κρίσεων που προκύπτουν. Η ενεργοποίηση του Κέντρου Επιχειρήσεων για το συντονισμό των αποστολών στο κέρας της Αφρικής αποτελεί αναμφισβήτητα το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δυνατότητας σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων. Ωστόσο αυτό το κέντρο δεν είναι μόνιμο, ούτε αποτελεί κεντρικό σημείο σχεδιασμού και διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ η στελέχωσή του είναι ακόμα ανεπαρκής. Η ίδρυση ενός επιχειρησιακού στρατηγίου είναι μια αναγκαιότητα που πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Γι' αυτό το λόγο θα δώσω ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το ζήτημα. Όσο αφορά στις δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τη δυνητική συνεισφορά των EU Battle Groups στο μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών στην ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας και στην πρόθεση της πολυεθνικής συνεργασίας. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι ως σήμερα δεν έχει αναπτυχθεί κανένα EU Battle Group, αν και θα μπορούσε να αποτελέσει δύναμη πρώτης εισόδου σε αρκετές περιπτώσεις, αποδεικνύει τις δομικές αδυναμίες στο μηχανισμό λήψης των αποφάσεων, αλλά και στη χρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων. Ακόμα και ο αναθεωρημένος μηχανισμός Ατένα δεν λαμβάνει επαρκώς τις ιδιαιτερότητες των EU Battle Groups και πρέπει να προσαρμοστεί περαιτέρω, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των κοινών δαπανών και να διασφαλιστεί ο δικαιότερος επιμερισμός της επιβάρυνσης των δαπανών στις διάφορες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Άρα χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία, και μεγαλύτερη ταχύτητα στην κινητοποίηση των κονδυλίων, τροποποιώντας κατάλληλα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Σε αυτό το σημείο επόψη των συναδέλφων θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες. Είναι προφανές κύριοι συνάδελφοι ότι το τωρινό πλαίσιο δεν λειτουργεί. Πρέπει να αναζητήσουμε όλους τους πιθανούς τρόπους για να υπερβούμε τη σημερινή κατάσταση. Τρίτον, πέρα από τις δομές της Ένωσης υπάρχει ένα σημαντικός αριθμός πρωτοβουλειών που έχουν αναλυφθεί από τα κράτη-μέλη, άλλοτε σε διμερή βάση, άλλοτε μέσω συμμετοχών σε ευρύτερους πολυεθνικούς σχηματισμούς και χρειάζεται να συντονίσουμε αυτές τις δράσεις υπό την αιγίδα ενός συνολικού σχεδιασμού και όχι να τις περιορίσουμε. Στόχος μας πρέπει να είναι η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των υπαρχουσών πρωτοβουλειών ανεξάρτητα από το πλαίσιο που αυτά επιχειρούν. Είτε είναι Ένωση, είτε είναι ΝΑΤΟ. Τέταρτον, πρέπει να αναπτύξουμε δομές και ικανότητες για να αντιμετωπιστούν οι σημερινές αδυναμίες. Άρα θέλει μια πιο διαρθρωμένη προσέγγιση, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι στρατιωτικές αερομεταφορές, τα ελικόπτερα, η ιατρική βοήθεια, τα κράτη-μέλη πρέπει να προωθήσουν συστηματικές αναθεωρήσεις στους τομείς της ασφάλειας και άμυνας με βάση εναρμονισμένα κριτήρια. Σε αυτό το πεδίο η συνεκμετάλλευση και ο επιμερισμός των ικανοτήτων pooling and sharing δεν αποτελεί επιλογή αλλά επίγουσα αναγκαιότητα πλέον. Για την επίτευξη αυτού του στόχου καθοριστική θα είναι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενεργονίσουν τους αμυντικούς σχεδιασμούς σύμφωνα με το Capability Development Plan. Υπάρχουν δε ήδη σημαντικά παραδείγματα που αποδεικνύουν τα σημαντικά περιθώρια επίτευξης συνεργειών και οικονομιών κλίμακος, τα οποία οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε. Παραδείγματο χάρη η κοινή ιδιοκτησία κάποιων ακριβών μέσων και ικανοτήτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μη στρατιωτικές χρήσεις είναι μια επιλογή που πρέπει να προωθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, στρέφοντας το βλέμμα προς το μέλλον, θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες συνεργασίας, συντονισμού και κοινών δράσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ενισχύσουμε και την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, της εξειδίκευσης και των κοινών ασκήσεων στην Ευρώπη η επιτυχία του προγράμματος Helicopter Training Program είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να αναδειχθεί και να συνεχιστεί και σε άλλους τομείς. Τελειώνοντας την παρουσίαση, θέλω να σταθώ στο τμήμα της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας. Η συνθήκη της Λισαβόνας εισάγει μια θεσμική καινοτομία που δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί. Γνωρίζω τις έντονες συζητήσεις που γίνονται στο Συμβούλιο επί του θέματος καθώς και το γεγονός ότι δεν υπάρχει ισχυρή πλειοψηφία για το πώς θα έπρεπε αυτό να προχωρήσει. Πιστεύω όμως ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο ένας ορισμός θα ήταν χρήσιμος επί του παρόντος. Είμαι όμως βέβαιη ότι θα πρέπει να βρεθεί κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στη θέσπιση πολύ αυστηρών κριτηρίων που θα λειτουργούν ως αντικίνητρα στη συμμετοχή των κρατών μελών και τις πολύ χαλαρές δεσμεύσεις που θα προσφέρουν ελάχιστη προσθεμένη αξία στην προσπάθεια οικοδόμησης μιας ισχυρής πολιτικής άμυνας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θέλω να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων. On behalf of Mr. Ο κύριος Πάσκου από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζετε σίγουρα ότι η προσέγγιση της κυρίας Γιαννάκου που παρουσιάζει καταρχήν τα έγγραφα πλαισίου είναι σημαντική γιατί όταν μπαίνουμε στις λεπτομέρειες θα πρέπει καταρχήν να ξέρουμε ποιο είναι το γενικό πλαίσιο. Νομίζω ότι η κυρία Γιαννάκου επίσης το έγγραφό της Εργασίας αναφέρει το γεγονός ότι η Ευρώπη δημιουργεί τώρα μια σωρία εργαλείων, αλλά όταν πρόκειται για τη χρήση αυτών των εργαλείων δεν τα χρησιμοποιεί. Μόνο με αυτοσχεδιασμούς λειτουργεί. Και το ερώτημα είναι γιατί προετοιμαζόμαστε για τη δημιουργία όλων αυτών των μέσων εάν δεν τα χρησιμοποιούμε. Εκεί πρέπει να δώσουμε λοιπόν έμφαση. Εκεί θα πρέπει να μετατρέψουμε τα λόγια σε δράσεις. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή εμοραγεί σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική δύναμη. Ξέρετε ότι κάποια στοιχεία που ήταν το, το βασικό χαρακτηριστικό της ισχύω μας έχουν χαθεί και επίσης με ναι, το τέλος πολλών επιχειρήσεων έχει μειωθεί πάρα πολύ η στρατιωτική ικανότητα και μέσα στο ΝΑΤΟ υπάρχει αυτή η μορφή προβληματισμού για το πώς θα μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε αυτή την εμπειρία η οποία έχει χαθεί και μόνο με ασκήσεις μπορεί να ανακτηθεί. Υπάρχει το θέμα του προϋπολογισμού στο ΝΑΤΟ προβλέπεται και μια διάσκεψη κορυφής για αυτό το θέμα της αναστολής της περικοπής των εθνικών προϋπολογισμών, στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Γκόμες πριν από μια ώρα, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι ακόμα είναι το γεγονός ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε, η οποία στο παρελθόν καλύπτε το 70% της ικανότητας του ΝΑΤΟ, έχει φτάσει να είναι το 80, το 85% και τώρα οι νομές Πολιτείες έχουν πει ότι θα το περικόψουν αυτό στο 50%. Και επομένως εμείς θα πρέπει να καλύψουμε τη διαφορά. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα πρέπει να περιληθούν σε αυτό το πλαίσιο και επομένως είναι απαραίτητο να έχουμε μια προβληματική για τα θέματα αυτά. Αλλά αν συνεχίσουν αυτές οι καταστάσεις θα πρέπει να διαχειριστούμε την, την σπάνιδα των ικανοτήτων μας. Δεν θα μείνει τίποτα να θέσουμε από κοινού. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να κρούσει τον κόνδωνα του κινδύνου γιατί έχουμε φτάσει τον πάτο του βαρελιού. Αν δεν θέλουμε να θέσουμε σε δραστική αμφισβήτηση την ασφάλειά μας, τότε πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε καλύτερα για όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Για την άλλη τώρα. Ναι, όπως είπαμε και για το σχέδιο κειμένο, συμφωνούμε με την ανάλυση της κατάστασης, αλλά δεν συμφωνώ όσον αφορά τι προοπτικέ για το μέλλον, γιατί για πρώτη φορά έχουμε αναλάβει κάποιον, έχει αναλάβει κάποιο την έκθεση, μάλλον που αντιμετωπίζει από αυτή την, την πολιτική οπτική γωνία τα πράγματα ακριβώ όπω μα τα παρουσιάσετε σήμερα. Πάντω, εν γέννη, συμφωνούμε με τι θέσει σα. Αλλά θα, αυτό που θέλω να σα τονίσω είναι τα εξή τρία. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε μια σοβαρή ανάλυση κατόπιν το Ελσίνκι, κατόπιν το Ελσίνκι, κατόπιν των όλων ε, επιχειρήσεων που έχουν γίνει. Έχουμε τα battle groups, το, το στρατηγείο, το, το στρατηγικό προσωπικό και αν προσπαθούμε να συγκροτήσουμε και άλλους φορείς, αυτό είναι κάτι σαν αιμορραγία θεσμική. Το θέμα είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτά που ήδη έχουμε, διότι νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Έχουμε τα battle groups, έχουμε το Europe Corps, αλλά για κοιτάξτε τι έγινε στο Μαλί. Θα θέλαμε να υπάρχουν και εθνικέ ενόπλε δυνάμει από την αρχή. Επίση, θα πρέπει ε, όλα αυτά τα ερωτηματικά να απαντηθούν. Αφού έχουμε κάτι, κάτι θεσμικά, γιατί δεν είμαστε προετοιμασμένοι, δεν είμαστε πρόθυμοι να το χρησιμοποιήσουμε και μετά τις συγκρούσεις. Ναι, να υπάρχει κάτι τέτοιο θεσμικά. Όμως, είναι δυνατόν να πληρώνουμε κάτι που δεν χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό είναι το δεύτερο ερωτηματικό που αναδύεται. Επίσης, Θα συνεργαστούμε, είναι πάρα πολύ ελαστική η προσέγγισή σας και πάρα πολύ αναγκαία διότι ενδεχομένως έχουμε αποφύγει να χρησιμοποιήσουμε την ξύλινη γλώσσα όπως γίνεται πολλές φορές αλλά όπως είπατε θα πρέπει η ευκαιρία να γίνει μια κρίση. Να είμαστε ρεαλιστές και τελικά κάτι να βγει από όλα αυτά όσον αφορά την κοινή πολιτική μας και την άμυνά μας. Συμπαθάτε με, αλλά έχω με κρυωμένη. Κυρία Κρόμπεργκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. I think there's a definition problem. Εδώ έχουμε πρόβλημα ορισμού. Για κοιτάξτε τον τίτλο και μετά. Μετά που μιλάμε για τις δομές, μετά μιλάμε για επιχειρήσεις και μετά μιλάμε για δυνατότητες, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες διακρίσεις σαφείς. Όσον αφορά τα battle groups, δεν αποκλείω το ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ότι έχουν υπάρξει περιπτώσει κατά τι οποίε θα μπορούσαν ή θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Αλλά νομίζω ότι για το στρατό και για τα οπλικά συστήματα το πιο ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι να μην χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν. Εκταμείβονται πάρα πολλά για όπλα στην Ευρώπη που δεν χρησιμοποιούνται, δεν αναλώνονται. Ή τέλο πάντων για όπλα που δεν χρησιμοποιούνται και άλλα. Άρα θα πρέπει να είμαστε πιο κοδηματικοί όσον αφορά τα battle groups που χρησιμοποιείτε Εμεί στην Φιλανδία, ε, όταν ε, εγκρίναμε τα battle groups, θεωρήσαμε ότι το γεγονό ότι υπάρχουν ε, δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο για την ενεργοποίησή του, χρησιμοποίησή του. Πέραν του τώρα, νομίζω ότι το επιχειρησιακό στρατηγείο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα και ότι και για κάποιες αυτόνομες επιχειρήσεις είναι κάτι το αναγκαίο και νομίζω ότι κάποια από τα υπάρχοντα κέντρα μπορούν να συγχωνευτούν τέλος για το pooling and sharing. Τα συζητάμε, τα ξανασυζητάμε, αλλά δεν προχωράμε και πάρα πολύ, αυτό είναι πρόβλημα. Και ακριβώς με δεδομένο ότι οι χώρες μέλη βάζουν τα λεφτά, χρειάζεται τελικά κάποιο είδου διαφορετική δομή για να προωθηθεί το pooling sharing και να μετεξελιχθούν και αν μετεξελιχθούν πώς θα γίνουν Turnbull έτσι έτσι δεν ονομάζεται Κάμπελ, α, Κάμπελ, Κάμπελ Κάμπελ, κυρία Πρόεδρε Ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ φοβάμαι ότι είμαι εντελώ αντίθετο με την κατεύθυνση που παίρνει αυτή η έκθεση. Δεν θα σα εκπλήξει αυτό και με ανησυχεί και η γλώσσα που χρησιμοποιεί. Νομίζω ότι το κατέστη σαφέ ε, ο στρατηγό προηγουμένω είπε ότι οι στρατιωτικές δυνάμει ανήκουν στα κράτη-μέλη και εδώ γίνεται αναφορά σε ευρωπαϊκέ ενοπλέ δυνάμει, σε ειδικέ ευρωπαϊκές δυνάμεις, χρήση στον ε, στρατιωτικών της ε, δυνατοτήτων, μα ποιανού είναι αυτές οι ένοπλες δυνάμεις, είναι των κρατών μελών, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει διαφορά. Μιλάμε για ζήτημα εθνικής κυριαρχίας και με ανησυχεί ιδιαίτερα το θέμα των battle groups. Έχω επισκεφτεί κάποια τέτοια battle groups στο Ηνωμένο Βασίλειο και Αναφέρεται ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ ευρωπαϊκά battle groups. Δηλαδή τι, θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε πόλεμο. Δεν είμαι, ξέρετε, υπερβολικά ευαίσθητος. Εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο είμαστε πολύ σοβαροί σε ό,τι αφορά τις ευθύνες μας στο Αφγανιστάν και ούτω καθεξής, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να αναφέρεται ότι μπορεί κάποιο άλλο να αποφασίζει για τι δικέ μα ε, ένοπλε δυνάμει. Ε, με ανησυχεί πάρα πολύ η έκθεση αυτή και θα την καταψηφίσω πολύ φοβάμαι. Thank you too. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τη διαφορά των ε, απόψεων που εκφράστηκε, λέει η πρόεδρο. Η κυρία Γιαννάκου, θέλετε να απαντήσετε στι παρεμβάσει αυτέ για να ολοκληρώσουμε μετά. Βεβαίω, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ του συναδέλφου εσά. Ε, τον ε, κύριο Πασκού, ε, την κυρία Κρόμπεργκ αλλά και τον κύριο Κάμελ για τις απόψεις που εκφράστηκαν. Καταρχήν, κύριοι συνάδελφοι, έχουμε μια δεδομένη πραγματικότητα. Η συνθήκη της Λισαβόνας δημιουργεί δομές. Φυσικά οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή ανήκουν και κατευθύνονται στα κράτη-μέλη. Αλλά τα κράτη-μέλη είναι αυτά που έχουν δημιουργήσει την Ένωση. Η οποία είναι μια ένωση συνδεδεμένη σε τέτοιο βαθμό που αποφασίζει στο 80% των αποφάσεων ε, στην πραγματικότητα συντονίζεται. Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι το ότι έχει κανείς στρατιωτικές δυνάμεις και δομές δεν σημαίνει σώνει και καλά ότι θα γίνει πόλεμος και θα τις χρησιμοποιήσει. Αλλά πρέπει να τις έχει. Για να έχει αυτή τη δυνατότητα. Το ίδιο κάνουν και τα κράτη-μέλη. Δηλαδή θέλω να πω στον κύριο Κάμελ ότι οι Βρετανικές ε, στρατιωτικές δυνάμεις τι κάνουν. Γιατί εκπαιδεύονται, είναι συνεχώς σε πόλεμο. Όχι. Υπάρχουν όμως. Και η συνθήκη της Λισαβόνας ε, γνωρίζω καλά ότι έχει εγκριθεί και από τη χώρα του. Επομένω δεν υφίσταται θέμα να έχει συμβεί κάτι χωρίς μια χώρα να το ξέρει ή να μην υπάρχει εθνική κυριαρχία. Εδώ λέμε ότι έχουμε τις δομές, έχουμε τους θεσμούς και δεν τους χρησιμοποιούμε όπως πρέπει. Και ταυτόχρονα εμφανίζεται μια δικαιολογία ότι υπήρξε η μείωση των αμυντικών δαπανών. Ναι, υπήρξε μείωση σε όλες τις χώρες. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα με συντονισμό και συνεργασία με πολύ λιγότερα χρήματα να κάνουμε πολύ περισσότερα και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που έκανε ο κύριος Πασκού αλλά και εσείς ε, κυρία Πρόεδρε τι να τα κάνουμε τα μέσα όπως είπατε και τους θεσμούς αν δεν τους χρησιμοποιούμε. Γιατί να έχουμε κόστος. Εγώ πριν α, ε, ε, αρχίσω να, να δημιουργώ την έκθεση συναντήθηκα και με τον ε, ε, στρατηγό Βανός ο οποίος ήρθε εδώ σήμερα και συζητήσαμε και η δική τους άποψη είναι επίσης ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα πιο συντονισμένα παραδείγματος χάρη πιο συντονισμένα πράγματα γίνανε στο κέρας της Αφρικής αν και δεν είναι τέλειο το σύστημα από ανθρώπους που ήδη υπάρχουν από δομές που ήδη υπάρχουν από τρόπους να υπάρξει κοινή εκπαίδευση. Άλλωστε θέλω να πω στους συναδέλφους ότι παραδείγματο χάρη κοινέ ε, ασκήσεις και κοινή εκπαίδευση υπήρχε πολύ πριν δημιουργηθεί η, ακόμη η ενιαία πράξη μεταξύ των κρατών διότι υπήρχαν διμερείς συνεργασίες ούτως ή άλλως δηλαδή ζούμε σε μια ε, κατάσταση πολυεπίπεδης συνεργασίας Άρα δεν φέρνουμε τίποτα το καινοφανές. Εγώ θα λάβω υπόψη μου όλα όσα ελέγχθησαν. Ε, φυσικά δεν μπορώ να λάβω υπόψη μου την άποψη του κυρίου Κάμελ ότι ε, θα πρέπει να είμαστε εναντίον αυτής της προσπάθειας. Το αντίθετο, αλλά τον ευχαριστώ έστω για την αντίθετη απόφασή του και θα λάβω υπόψη μου τις παρατηρήσεις του κυρίου Πασκού, ο οποίος άλλωστε υπήρξε και υπουργό Εθνικής Άμυνας και γνωρίζει βαθύτερα τα ζητήματα και έχουμε συνεργαστεί και πάλι, εσάς κυρία Πρόεδρε και της κυρίας Κρόμπερ και όλων των συναδέλφων που θα θελήσουν να κάνουν παρατηρήσεις και να στείλουν γραπτός κάποια σημειώματα τα οποία θα μπορούσαν να συνεισφέρουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η συζήτηση για την έκθεση θα γίνει στις 9 Μαρτίου. Κλείνω τη συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση στις 7 Μαρτίου στις 9 το πρωί.